Chers collègues, si vous voulez bien rejoindre... Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε οι επισκέπτες το ίδιο στο βάθος της αίθουσας. Απενεργοποιήστε παρακαλώ τα κινητά σας. Σταματήστε τις ιδιωτικές συνομιλίες για να μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Bien. J'ouvre la séance. Au point 1, nous... Άρχεται η συνεδρίαση. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσια διάταξης. Μια και δεν έχω λάβει σχόλια, προτείνω να την υιοθετήσουμε μετάβλητη. Σημείο 2. Πρακτικά της συνεδρίασης της Δευτέρας και 3ης Σεπτεμβρίου. Τα έχετε λάβει, δεν έχετε στείλει παρατηρήσεις, αλλά τα θεωρώ συγκεκριμένα. Σημείο 3. σεπτεμβριου τα εχετε λαβει δεν εχετε στειλει παρατηρησεις αλλα τα θεωρω συγκεκριμενα σημειο 3 ανακοινωσεις της Προέδρου. Δύο ανακοινώσεις έχω. Καταρχήν, μην ξεχνάτε ότι η αυριανή μας συνεδρίαση ακυρώθηκε και να σας επισημάνω ότι βρίσκεται κοντά μας μια αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεταφορών. Στο σημείο 4 σας προτείνω κοινή συζήτηση των σημείων 4 και 5 γιατί και τα δύο αφορούν το ίδιο θέμα, είναι αλληλένδετα. Το πρώτο αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη και το δεύτερο το κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και κοινωνική αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα Progress δηλαδή. Και για τα δύο θέματα η συγγήτρια είναι η κυρία Κίνκα Γκέντς. Χωρίς άλλη χρονοτριβή θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Αν δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και αίθουσα ακρόασης που είναι, βρίσκεται ακριβώς δίπλα είναι η 1G2. Επίσης η συνεδρίαση να μεταδίδεται στο web streaming. Οπότε ό,τι λέτε και κάνετε αναμεταδίδεται. Η κυρία Κίνκα Γκέντς, σας ευχαριστώ. Χάρηκα ιδιαιτέρως ε, ότι υπάρχει υποστήριξη ε, και της G20 με δήλωσή της για το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Πέραν όμω ε, τη συμφωνία των G20, έχουμε να εγκρίνουμε και κάποιε τροπολογίε. Συναντήθηκα με τον Επιτροπό Σπίτλα, με τη Σουηδική Προεδρία, τι διάφορε επιτροπέ. Είχα διαβουλεύσει και με μη κυβερνητικέ οργανώσει που ενεργοποιούνται στο θέμα αυτό και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και από ό,τι βλέπω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να δέχεται τη νέα δημοσιονομική γραμμή, την αυτοτελή δημοσιονομική γραμμή, που ήταν ένα από τα βασικά θέματα διαφιλονικίας πέραν των τροπολογιών. Και το επιχείρημά μας ήταν ότι η φιλοσοφία του προγράμματος ε, αυτού είναι κάπως διαφορετική από τη φιλοσοφία του προγράμματος Progress. Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει τα πλέον ευάλωτα άτομα και τις πιο μειονεκτικές κατηγορίες αλλά υπάρχει διαφορετικό είδος συνδυασμού πόρων των δύο προγραμμάτων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοτελή δημοσιονομική γραμμή για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Ελπίζω να εισακουστεί το έτοιμά μας και να το δεχτεί τελικά και να το εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έγιναν προτάσεις ε, για καλύτερο ορισμό και οριοθέτηση της μικροχρηματοδότησης, της μικρής ε, επιχείρησης ε, και του δικαιούχου. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, εκτός από τη δική μας πρόταση για αυτοτελή, δημοσιονομική γραμμή και νέα κονδύλια, προτάθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια το ποσό, δηλαδή από 100 να γίνει 150 εκατομμύρια. Και το ΕΛΚ προτείνει, προτείνει 40 εκατομμύρια για το 2010 που θα είναι το πρώτο έτος λειτουργίας. Και η Επιτροπή Περιφερειών πρότεινε να διαδραματίζουν ρόλο στο πρόγραμμα και η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ε, παρακολούθηση. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Να κάνω μια σύντομη επισκόπηση των τροπολογιών καταρχήν. Ε, ένα προβληματικό θέμα ήταν ε, ο ορισμός του ε, πελάτη, των ε, δυνάμει πελατών. Και αντί να έχουμε εξαντλητική απαρίθμηση των διαφόρων κατηγοριών πελατών, υπευλήθη μια πρόταση που είναι αρκετά αδόκιμη. Να πούμε δηλαδή, όσοι αποκλείονται από την συμβατική αγορά πιστώσεων, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος, να επιτρέψει πρόσβαση σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στι εμπορικές ή συμβατικέ πιστώσεις. Και ελπίζουμε μετά το πρόγραμμα αυτό να εξασφαλιστεί και η πρόσβασή του στη συμβατική αγορά πιστώσεων. Δεχόμαστε λοιπόν τον ορισμό που λέει ότι η επίδοξη πελάτες είναι αυτοί που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και που έχουν δυσκολία ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί τη χρυσή τομή νομίζω μεταξύ των διαφόρων προτάσεων. Και αν χρειαστούν διευκρινήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Η πρόταση της Επιτροπής Περιφερειών έλεγε ότι κάποιες ε, μη εμπορικές ε, χρηματοπιστωτικές ε, οργανώσεις που δίνουν μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να υποστηριχθούν. Και τονίστηκε η σημασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ε, προσπάθεια αυτή για τη στήριξη αυτών των ε, παρόχων μικροχρηματοδοτήσεων. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και στην ε, ατομική καθοδήγηση των πιθανών πελατών η στήριξη δηλαδή της μικροχρηματοδότησης να συνοδεύεται από τομική καθοδήγηση και κατάρτιση ώστε να μπορέσει ο πελάτης να αναπτύξει ένα βιώσιμο πρόγραμμα. Και μετά από διαβουλεύσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις θέλουμε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ότι ο ε, με τα υπάρχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα καθώς και μέτρα κοινωνικής ε, στήριξης ε, χρειάζεται ο συντονισμός αυτός είναι απαραίτητος για να έχουμε την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Έγιναν κάποιες συζητήσεις για την ομάδα των πελατών των δικαιούχων και ε, υπευλήσαν πολλές προτάσεις για τον ορισμό των δικαιούχων των πελατών. Ζητήσαμε, επαναλαμβάνω, αυτοτελή δημοσιονομική γραμμή, νέο κονδύλιο και όχι μεταφορά κονδύλιων από το Progress. Ελπίζω να εγκριθεί αυτή η πρότασή μας για 150 τελικά εκατομμύρια. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συμπληρώσει με κονδύλια αυτό το ποσό. Δηλαδή, πρώτος ε, πάροχο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και ευελπιστούμε ότι και εμπορικές τράπεζε. Ε, θα συμβάλλουν στο πρόγραμμα ώστε να εμπλουτιστούν οι πόροι. Συζητήθηκε πώς θα εξασφαλίσουμε πρόσβαση όλων όσων χρειάζονται τέτοιου είδους στήριξη στο πρόγραμμα. Γι' αυτό και συντάξαμε μια τροπολογία που μιλά για στενή παρακολούθηση της διαδικασίας και τη χρήση των κονδυλίων που παρέχει το εχέγγυο ότι όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι δικαιούχοι, οι πιθανοί δικαιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια. Παρόλο που σε ορισμένε χώρε υπάρχει, υπάρχει τέτοιο σύστημα μικροπιστώσεων και μικροχρηματοδοτήσεων. Σε άλλε όμω χώρε δεν υπάρχει καμία τέτοια παράδοση, καμία τέτοια εμπειρία μικροχρηματοδοτήσεων ή μικροπιστώσεων. Γι' αυτό και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ ε, την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και να δούμε πώς γίνεται η διανομή των κονδυλίων, ώστε πραγματικά να φτάσουν τα κονδύλια αυτά σε όλους τους ε, ε, επίδοξου πελάτε ή του δικαιούχου που τα χρειάζονται. Μία άλλη τροπολογία προβλέπει ότι στην ετήσια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει προσπελασιμότητα του μέσου αυτού σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Κάτι άλλο που εξετάσαμε αφορά το πρόγραμμα Progress και λέμε ότι δεν συμφωνούμε με την πρόταση να συνδυαστεί αυτή η δημοσιονομική γραμμή ε, με το πρόγραμμα Progress ή να αφαιρεθεί το κονδύλιο αυτό από το πρόγραμμα Progress. Γιατί το είχαμε πει ήδη από την αρχή, δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση να γίνει μεταφορά κονδυλίων από το Progress. Και εμείς αρχικά είχαμε προτείνει αύξηση της δημοσιονομικής γραμμής του Progress. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφασίσει αφαίρεση των κονδυλίων αυτών από διάφορα τμήματα του Progress ουσιαστικά ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε σε τέτοιου χαλεπού καιρού, με ζούσει τη κρίση και με δεινή κοινωνική κατάσταση σε πολλέ χώρε, ήταν πολύ λάθο μήνυμα να στείλουμε μια περικοπή των κονδυλίων του Progress και άρα μια αποδυνάμωση της υποστήριξης. Εμείς το αντίθετο θέλουμε να πούμε ότι ενισχύουμε την υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται. Ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκέντς. Η ε, κυρία Λίν και μετά ο κύριος Έλμερ. Σύνομα δύο σημεία για τους αυτοαπασχολούμενους. Χαίρομαι που συμπεριελήφθησαν στη συγκεκριμένη έκθεση. Στο 2β για τους ανθρώπους με συγκεκριμένα προβλήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νέοι. Γιατί πάρα πολύ συχνά είναι σαφές ότι οι ηλικιωμένοι απολύονται και το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους νεότερους που έχουν δυσκολίες σε σχέση με τα οικονομικά τους. Για το progress τώρα, μια ερώτηση. Τίνω να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε. Ο προϋπολογισμός του Progress εν πωλής έχει δαπανηθεί, έχει ε, καταναλωθεί. Και υπάρχουν κάποια άλλα ταμεία τα οποία ε, δυστυχώς δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Και εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει, ίσως θα πρέπει να υπάρξει και για το πρόβλημα της μικροχρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των μικρών και μικρότερων επιχειρήσεων, ένα, μια ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλμερ ανησυχώ λίγο από αυτά τα οποία ακούγονται εδώ γύρω. Όλοι γνωρίζουμε ότι βιώνουμε μια σκληρή οικονομική κρίση και η απάντησή μας στην κρίση αυτή είναι ότι επειδή υπάρχει θα πρέπει φυσικά να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα, να ξοδεύουμε περισσότερες πιστώσεις. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Νομίζω ότι στα περισσότερα και στο δικό μου οι κυβερνήσεις λέγονται ότι ε, μια και βρισκόμαστε στα πλαίσια μια οικονομική κρίση πρέπει να ξοδεύουμε λιγότερα. Ακόμα και οι εργατικοί αποφάσισαν ότι αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι πολλοί από εμά βρίσκουν λίγο περίεργη τη στάση αυτή. Όταν οι οικονομίε μειώνουν του προπολογισμού του. προσπαθούμε εμεί να βρούμε λύσει για να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα. Παράλογο. Έχουμε επίσης και κάποια προβλήματα ορισμών Ποιοι είναι οι λεγόμενοι πελάτες, χρήστες. Προφανώς ε, πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις και γι' αυτό θα παίρνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα. Θα υπάρχουν πολλοί που θα ωφεληθούν, οπότε το κόστος διαχείρισης θα είναι τεράστιο. Κανένας δεν μίλησε για το κόστος της διαχείρισης του προγράμματος αυτού και πολύ φοβάμαι ότι ένα μεγάλο τμήμα του διαθέσιμου ποσού θα χαθεί εκεί. Τώρα για την επιλογή ε, των πελατών σε εισαγωγικά, αυτών που θα ωφεληθούν εν πάση περιπτώσει, η εισηγήτρια είπε ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε όλους τους δυνατούς χρήστες, πελάτες. Και η κυρία Λίν ε, είπε ακόμα περισσότερο ότι και τους νέους και τους ηλικιωμένους θα πρέπει να συμπεριλάβουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτά τα λίγα χρήματα θα τα μοιράσουμε σε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων ε, και δεν νομίζω ότι θα κερδίσει κανείς κάτι από αυτό. Και προφανώς δεν θα πετύχουμε τον στόχο αυτό να φτάσουμε δηλαδή σε όλους τους πιθανούς εισαγωγικά πελάτες. Λέμε ότι το πρόγραμμά μας είναι να στοχεύσουμε αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εμπορικά ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι τα χρήματα για τα οποία συζητάμε είναι πραγματικά τίποτα σε σχέση με την μεγάλη μείωση στον τομέα της δανειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό λοιπόν το άγχος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις ε, επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις πιο καινούργιες πρόσφατες επιχειρήσεις χωρίς παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πολύ προσεκτική επιλογή ε, για αυτούς οι οποίοι θα ωφεληθούν. Και αν το κάνουμε αυτό βέβαια θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ η τόσο προσφυλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδος του μέσου. Πρέπει λοιπόν ό,τι αποφάσεις να πάρουμε να τις πάρουμε με ουδέτερο τρόπο, να μην ευνοήσουμε κανέναν και να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να μειώσουμε το φορολογικό βάρος να μειώσουμε επίσης και τις ρυθμίσεις και τις νομοθετικές δεσμεύσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει βήματα προς τα πίσω. Και όχι το να δίνουμε λίγα χρήματα δεξιά και αριστερά σε κάποιους οι οποίοι μπορεί και να τα χρειάζονται, μπορεί και όχι. Thank you uh, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε πιστεύω όλοι ότι η ανάγκη, η, η ανάγκη τώρα να ξεκινήσουν οι, τα προγράμματα αυτά των ε, μικροχρηματοδοτήσεων είναι αδύρυτη. Οι μηχανισμοί αυτοί των μικροπιστώσεων ε, μπορούν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες σε νέες ομάδες πολιτών και μάλιστα από διάφορα επίπεδα ή στρώματα της κοινωνίας και δεν νομίζω ότι είναι πάντα χρήσιμο να μιλούμε για συγκεκριμένα στρώματα. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να στρεφόμαστε προς τους νέους, αλλά και άλλοι πολλοί, ε, επί παραδείγματι εκείνοι που κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας τους ή που έχουν μείνει ανεργοί, θα πρέπει να αποτελούν στόχο μας. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουμε περισσότερο στην υπόθεση αυτή είναι σχετικά με την χρηματοδότηση του κονδυλίου αυτού. Άρα λοιπόν πρέπει η λύση που θα βρεθεί να είναι η καταλληλότερη έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Και έχουμε πολλά ζητήματα πιστεύω χρηματοοικονομικού τύπου που θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή μας. Επί παραδείγματι, το γιατί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει αυτή τη σημαντική δράση από τον προπολογισμό για την πρόοδο και πώς θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών κατά τρόπον ώστε τα ποσά που τελικά θα κατανεμηθούν να φτάσουν ε, στο επίπεδο των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης θα θέλω να ρωτήσω πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τα μη απορροφηθέντα κονδύλια. Ευχαριστώ η κυρία Μαρία Νάρκιν και μετά ο κύριος Τόμας Χέντελ. Κυρία Άρκιν Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ να υπάρχει μια ανεξάρτητη δημοσιονομική γραμμή, όπως είπε ο Γενικά από τους ψηφοφόρους μου οι παρατηρήσεις που ακούω πάντοτε είναι η δυνατότητα όχι μόνο της χρηματοδότησης αλλά της πρόσβασης στις μικροπιστώσεις είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στον Ευρωπαίο πολίτη. Και ναι, μπορεί να μην λύνει κάθε πρόβλημα αλλά πάντως αποτελεί τη σωστή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση το να κοιτάξουμε την ε, δυνατότητα πρόσβασης. Έχω πολλές επαφές εγώ στην ε, δική μου την ε, περιοχή με οργανώσεις, ε, μάλιστα και διεθνώς ε, ανεπτυγμένες, ε, με ανάπτυξη παραδείγματα στην Πολωνία, την Ιρλανδία, τη Βρετανία, τη Ρουμανία και άλλες, οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά ιδιαίτερα. Και όταν λέει ο συγητής ότι έχουν ανεπτυγμένο δίκτυο μικροπιστώσεων ορισμένε χώρε. Ναι, όντω μπορεί να ισχύει αυτό και νομίζω ότι από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα θα προκύψει ότι δεν υπάρχουν σε άλλε χώρε αντίστοιχα δίκτυα και ίσω μπορούμε να υποφεληθούμε από τι γνώσει που έχει να προσφέρει ο ένα τον άλλον. Αλλά πάντω υπάρχουν δίκτυα τουλάχιστον διεθνώς ανεπτυγμένα. Ε, και νομίζω ότι όταν πρόκειται να ξεκινήσει ε, εάν είναι να ξεκινήσει κάποιο προσδιορισμό ομάδων, θα πρέπει να επιτραπεί πρόσβαση στου πάντε. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρξει κανένα προσδιορισμό. Επίση, ε, πέραν τη μικροπίστωση, θα έπρεπε ίσω να αναφέρεται η έννοια των υπηρεσιών αποταμίευση, γιατί νομίζω ότι ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να καλύψουμε και το θέμα αυτό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πτυχή της ανάπτυξης ενεργητικού. Διότι το πρόβλημα που είχαμε πάντοτε με τις μικροπιστώσεις, ε, με ε, με γενικά με την πρόσβαση σε πιστώσεις, ήταν ότι κάποιος δεν, δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τις απαραίτητες εγγύησεις και γι' αυτό δεν μπορούσε να εξασφαλίσει πίστοση. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτή την πτυχή της παράλληλης αποταμίευσης ή της ε, συμπερίληψης τη αποταμίευσης. Επίσης, ε, ως ε, κάποια η οποία πρόκειται να υπερψηφίσει στο δημοψήφισμα για την συνθήκη της Λισαβόνας, θα ήθελα να σημειώσω παρεμπιπτόντως ότι πρόκειται για ζήτημα επικουρικότητας που θα έπρεπε να επαφευθεί στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος που χρησιμοποιείτε και την ε, αναμετάδοση της συνεδρίασής μας για να κάνετε και την εκστρατεία σας στη χώρα σας. Παρακαλώ, κύριος Χάντελ να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Χέντελ για την ακρίβεια. Από την ομάδα των Πρασίνων θα ήθελα ρητά να πω ότι υποστηρίζουμε την έκθεση της κυρίας Γκέρνς κατ' ουσίαν. Θα ήθελα ωστόσο να κάνω μία παρατήρηση μόνο. Ε, μία φράση που συχνά ακούμε στη Γερμανία, παροιμιακή φράση θα έλεγα, ότι όταν δεν φτάνει να μοιράσουμε σε όλους, εξοικονομούμε από τους φτωχούς. Και αυτό το λέω για κάποιους από τους ιδιαίτερα προτείνουμε λοιπόν την έκθεση αυτή να μην την απορροφήσουμε από τα κονδύλια του progress αλλά από άλλη ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Και κάτι ακόμη ότι μας λείπουν τα ποσά. Μπορεί να μην φτάνουν ενδεχομένως τα 150 εκατομμύρια 100% ή να μην φαίνονται πολύ γενναιόδωρα ποσά αλλά πάντως ίσως θα ήταν καλό να έχουμε υπόψη ότι το ότι το, ότι το γεγονός ότι το ποσό αυτό ιδιαίτερα είναι αφιερωμένο σε ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να ε, επωφεληθούν από άλλου τύπου πιστώσεις ή δανεισμό δεν είναι καλή λύση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αναφορά και πιστεύω ότι θα έπρεπε κατά τη διάρκεια ενός startup περιορισμένων ε, διαστάσεων εκκίνησης δραστηριότητας επιχειρηματικής να υπάρχει και κάποιο είδους ε, ανάδοχος αν θέλετε ή κάποιος ο οποίος θα φρόντιζε να βοηθήσει και να υποστηρίξει και με την τεχνογνωσία των ε, τον επιχειρηματία. Αυτό μαζί με τα προγράμματα START, start θα μπορούσε να λειτουργήσει και να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης, εκ παραλίλου δηλαδή. Και επίσης θα ήθελα να επαληθευθεί μέσα στην έκθεση της κυρίας ε, ένα σημείο στο κείμενο ή μάλλον δύο σημεία στο κείμενο που βρίσκω ότι δεν είναι πολύ σαφή και ίσως να οδηγήσουν σε αυθαιρεσίες στην τροπολογία υπαριθμών 8 καταρχάς έχασαν ή κινδυνεύουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την είσοδο ή επανείσοδο του στην αγορά εργασίας, πάλι στην τροπολογία 8, δυσκολίες για την είσοδο ή επανείσοδο και στην 9 αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Και οι δύο διατυπώσεις είναι υπερβολικά αόριστες. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, ενδεχομένω λαμβάνοντα και κάποιε προτάσει από πραγματογνώμονε, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με τα κριτήρια που θα ορίσουμε. Επίση, θα ήθελα να καταθέσω και δύο τροπολογίες για συμπλήρωμα ε, του κειμένου εκ μέρους της ομάδας μου, διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτές οι πιστώσεις να ε, αποσκοπούν και στην ενίσχυση της ε, οικονομίας, της λειτουργίας οικονομίας πρώτον και δεύτερον ότι το πρόγραμμα δεν πρόκειται, δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί ή μάλλον να τύχει καταχρήσεων κατά τρόπον ώστε να ανατραπούν οι συνθήκες κοινωνικής προστασία ή το κοινωνικό κράτος στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ελίζα Γιακοντσάρη και μετά η κυρία Ελισαμπέτ Μόγα. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ιδέα και χρήζει υποστήριξη. Το θέμα είναι πώς θα την εφαρμόσουμε και στην πράξη. Γιατί αυτή είναι η μοφή προς τα κοινοτικά προγράμματα ότι ήταν υπερβολικά δύσχρηστα και περίπλοκα. Πολλά πανεπιστήμια και μη κυβερνητικέ οργανώσει ήδη έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχουν παρετηθεί από τη χρήση των κοινοτικών προγραμμάτων, ακριβώ γιατί χρειάζεται να προσφύγουν σε επαγγελματίε για να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα. Και η προσπάθεια και το γραφειοκρατικό άχθος που συνδέεται με τα κοινοτικά προγράμματα είναι ενυπόφορα γιατί μπορεί να τα δημιουργήσουν τα κράτη-μέλη, αλλά συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη γραφειοκρατία. Έτσι, πολλοί προτιμούν να παρετηθούν, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, παρά να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλούμε για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια δινή κατάσταση. Είναι άνεργοι ή κοινωνικά αποκλεισμένοι, βρίσκονται σε μειονεκτικές ομάδες. Φροντίσαμε να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος και το διοικητικό κόστος ώστε να μπορεί κανείς να έχει όντως εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων και μικροπιστώσεων. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να είστε όρθιοι. Στη διπλανή αίθουσα, στην 1G2, έχει προβλεφθεί αίθουσα ακρόασης για τη συνεδρίαση αυτή. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και από εκεί. Ε, δεν είναι ακόμη έτοιμη μάλλον. Σε ένα δεκάλεπτο θα είναι έτοιμη. Οπότε όσοι είναι τώρα όρθιοι θα μπορούν να πάνε δίπλα για να καθίσουν. Η κυρία Ελιζαμπέτ Μογά και μετά η κυρία Πασκάλ Γκρούνη. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε καταρχήν ποιος είναι ο στόχος μας στο θέμα αυτό. Και στόχος μας είναι να επανέλθουν στην αγορά εργασίας ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί, δεν έχουν ενταχθεί ποτέ ή κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας. Και στόχος μας είναι μια αποτελεσματικότητα στο θέμα αυτό. Κατά την εφαρμογή ε, των μικροχρηματοδοτήσεων χρειαζόμαστε ένα λειτουργικό μηχανισμό ώστε να επιτρέπει την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας ή την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά κυρίως την επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και χρειάζονται μέτρα στήριξης. Μερικοί μίλησαν για ατομική καθοδήγηση, άλλοι μίλησαν για κατάρτιση. Πάντως χρειάζονται τέτοια συνοδευτικά μέτρα στήριξης πέραν των μικροχρηματοδοτήσεων που είναι εξίσου σημαντικά. Γιατί αυτή η την εισοδο στην αγορα εργασιας αλλα κυριως την επιτυχημενη εισοδο στην αγορα εργασιας γι αυτο και χρειαζονται μετρα στηριξης μερικοι μιλησαν για ατομικη καθοδηγηση αλλοι μιλησαν για καταρτιση παντως χρειαζονται τετοια συνοδευτικα μετρα στηριξης περαν των μικροχρωματοδοτησεων που ειναι εξισου σημαντικα γιατι αυτη η καθοδηγηση και η παρακολούθηση θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτού του μέσου. Και επιμένω σε αυτό, γιατί δεν θα ήθελα υπό το πρόσχημα ότι θεσπίζουμε ένα μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων να ευνοήσουμε κάποιους μηχανισμούς ε, κατάρτισης ε, αφιλεγόμενης ε, αποτελεσματικότητας ως προς τη διάρκεια τουλάχιστον, ως προς την αμεσότητά τους. Γι' αυτό και όσο καλές προθέσεις και αν έχουμε, αν ε, οι στόχοι μας ε, παρακολουθούν από τέτοιου είδους μηχανισμούς, ε, δεν θα υλοποιηθούν. Θέλουμε να ενισχύσουμε ένα είδος εθελοντικής καθοδήγησης και στήριξης που θα είναι το εχέγιο της αποτελεσματικότητας αυτού του μέσου. Δεν θα πρέπει να στηριχτούμε μόνο στο οικονομικό σκέλος της μικροχρηματοδοτήσης. Για να μπει κανείς αποτελεσματικά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας χρειάζεται και καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ κυρία Φυσικά και υποστηρίζω αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπέτ Μωρά. Προφανώς πρέπει να καλύψουμε την προσδοκία αυτή για μικροπιστώσεις για, τα, για τους πολίτες και τις εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα σε αυτή την περίοδο κρίσης. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τα κριτήρια για αυτές τις μικροπιστώσεις. Από ό,τι φαίνεται τα κριτήρια αυτά τα αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αν εμείς βάλουμε κατηγορίες νέοι, ηλικιωμένοι και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, τότε φοβάμαι ότι θα μειώσουμε την δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Κύριος Όρη, Τζάμπα Όρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχει ακουστεί επανειλημμένα ότι το μήνυμά μας είναι να δημιουργήσουμε πρώτο νέες θέσεις εργασίας αφού φυσικά συγκρατήσουμε τις υπάρχουσες. Εκεί βρίσκεται θα έλεγα ο πραγματικός στόχος της κίνησής μας και αυτό θα γίνει μέσω της ε, δημιουργίας μιας οικονομίας η οποία θα διευκολύνει και θα ευνοεί την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για να το πετύχουμε αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις λεγόμενες μικροεπιχειρήσεις και όταν λέω μικροεπιχειρήσεις αυτές οι οποίες είναι μικρότερες από το μέσο όρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις περισσότερες χώρες μας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να βοηθηθούν. Όπως για κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, οι δυσκολίες είναι θα έλεγα και στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλές. Εδώ και λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θα έλεγα κοινοβουλευτικής εντολής, έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από το λεγόμενο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ένα ταμείο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν καταναλώθηκε σε ικανοποιητικό ποσοστό, δεν απορροφήθηκε όπως λέμε με ικανοποιητικό τρόπο. Το θέμα είναι λοιπόν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να τα καταναλώνουμε διότι αλλιώς φοβάμαι ότι γινόμαστε αναξιόπιστοι. Το πρόγραμμα πλαίσιο αφορά ένα θα έλεγα μεσοπρόθεσμο χρόνο ε, από πενταετία μέχρι επτά χρόνια μάλλον και ακριβώς αυτό απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη ε, ικανότητα πρόβληψης έτσι ώστε οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Πρέπει όμως πριν από οτιδήποτε άλλο να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα τα οποία ζητάμε να διατεθούν θα είναι χρήματα, θα είναι πιστώσεις οι οποίες πράγματι θα απορροφηθούν. Μόνο τότε και εφόσον είμαστε σίγουροι μπορούμε να ζητήσουμε για επιπλέον πιστώσεις. γιατί ε, αλλιώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε απλά να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2010. Θα δούμε αν θα υπάρξει μια ξεχωριστή γραμμή για το μέσο αυτό της μικροχρηματοδότησης. Θα το διεκδικήσουμε. Αν θα το πετύχουμε σε αυτή τη φάση είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσω απάντηση. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά ότι η σλοβακική νομοθεσία σχετικά με την χρήση της ουγγρικής γλώσσας δεν έχει αλλάξει και γι' αυτό συνεχίζω να την ομιλώ. Ευχαριστώ κύριε Σκοφεράτη. Σεύτζο Κοφεράτη. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά φιλόδοξους στόχους αφιλόδοξη αλλά και εφικτή παρόλες τις δυσκολίες που φαίνεται να υπάρχουν. Όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το μέσο μικροχρηματοδότησης χρησιμεύσε για να παράσχει άμεση προστασία στους συμπολίτε μας που έχουν πρόβλημα να μπουν στην αγορά εργασίας και σε αυτούς οι οποίοι κινδύνευαν να χάσουν τη θέση απασχόλησης την οποία είχαν την παραγωγική τους δραστηριότητα εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να εισάγουμε και την έννοια της καινοτομίας έτσι ώστε να μετατραπεί αυτό το μέσο μικροχρηματοδότηση σε ένα ουσιαστικό μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε το μέσο αυτό και με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα στα πλαίσια των περιφερειακών και τοπικών ακόμα προγραμμάτων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σαφής αναφορά στα προγράμματα αναδιοργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας είτε για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας είτε για την προστασία και την περαιτέρω ανάπτυξη της βιοτεχνίας γενικότερα σε τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι που φύγεται σε τοπικό επίπεδο και γι' αυτό χρησιμοποιούν όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, τους ιδίους πόρους, προς εμπορικές αυστηρά διαστηριότητες με ό,τι αυτό σημαίνει. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι αυτή η οποία λειτουργεί θα έλεγα χρονικά πολύ πιο σύντομα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στρέψει κανείς την προσοχή του σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν σαν στόχο την παροχή συγκεκριμένων ποιοτικού επίπεδου υπηρεσιών ή και την παραγωγική πράγματι διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν το μέσο το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την έρευνα της καλύτερης ε, δυνατής δραστηριότητας στην οποία θα πρέπει να στραφούν αυτοί οι οποίοι έχουν δυσκολίες. Το θέμα δεν είναι να τους δώσουμε κάποια χρήματα για να αντικαταστήσουμε τα έσοδα τα οποία δεν έχουν άλλωστε στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά να είναι κάτι το οποίο συνδέεται με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στο μέλλον και να διαρκέσουν μία κάποια χρονική περίοδο. Δεν εννοώ υπερβατικά το θέμα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε στη διάθεσή μας νομίζω ένα μικρό βέβαια, αλλά σαφές μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Ο κύριος Μαν και μετά η κυρία Σόιτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Ρότζερ Χέλμερ ήταν εκείνο ο οποίο ήταν ο πιο επικριτικό εναντί αυτού του θέματος. Έλεγε ότι ε, πετάμε τα λεφτά από το παράθυρο σε μια εποχή όπου θα έπρεπε να είμαστε πιο οικονόμοι. Και τώρα μα λέτε ότι δεν δίνουμε τα χρήματα εκεί που πρέπει και ότι τα μοιράζουμε άκρητα. Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, όταν όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν τα χρήματα που τα έχουν ανάγκη, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα είχαν καμία άλλη ευκαιρία για να λάβουν πίστοση και σε αυτούς ακριβώς θα πρέπει να στοχεύσουμε να εξασφαλίσουμε την πίστοση. Και βέβαια ταυτόχρονα και να αναπτυχθούν θέσεις εργασίας. Βεβαίως, ναι, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος όταν επενδύουμε χρήματα να μην ξέρουμε τελικά τι προϊόν θα προκύψει, τι καρπό θα αποδώσουν. Και από την άλλη βεβαίω θα πρέπει να αποφύγουμε να μην υπάρχουν διπλές και τριπλές χρηματοδοτήσεις. Αλλά νομίζω ότι με μια απλή, ξεκάθαρη ερμηνεία μπορούμε να έχουμε ε, απλή εικόνα των κριτηρίων που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε. Είναι κάτι άλλο το οποίο έχουμε δει ήδη στη Γερμανία. Εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται μεγάλοι χορηγοί, κύριοι χορηγοί, που κάνουν το σύστημα να λειτουργεί δηλαδή και τα γρανάζια του, να μην είναι και οι ουσιαστικοί παράγοντες που ανατρέπουν μια κατάσταση. Δηλαδή τα μικρά κονδύλια να έχουν πολύ περισσότερη αποδοτικότητα από τα μεγάλα. Γιατί βεβαίως χρειαζόμαστε την υποστήριξη και των μεγάλων επιχειρήσεων ή ξέρω εγώ, την ε, ε, μέτρα τα οποία δεν θα κάνουν κακό στις μεγάλες επιχειρήσεις. Βεβαίως χρειαζόμαστε την υποστήριξη των μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ασφαλώς πρέπει να φροντίσουμε οι πιο αδύναμες ομάδες, οι πολύ αδύναμες ομάδες να έχουν μια πραγματική ουσιαστική ευκαιρία. Ευκαιρία η οποία ταυτόχρονα είναι συνειφασμένη και με την ευθύνη. Γιατί αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να προκύπτουν θέσει εργασία. Πρέπει να υπάρχει αυτό το κριτήριο. Η πρόσβαση λοιπόν και η αξιοποίηση κονδυλίων που θα ε, εξυπηρετούν πραγματικά το στόχο για τον οποίο έχουν διατεθεί. Και νομίζω ότι και στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ κυρία Σρόντερ. Ευχαριστώ. Φτάσαμε κάποια καθυστέρηση στην ε, συνεδρίες χαστήσει όμως ε, να παρακολουθήσουν για μένα την συζήτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό αυτών των μικροπιστώσεων. Ξέρετε ότι ε, έχω αρκετή εμπειρία από, τα, από τους μηχανισμούς αυτούς και από τα περιφερειακά κονδύλια και από τα περιφερειακά ταμεία και από αντίστοιχου τέτοιου μηχανισμού. Και γι' αυτό, με την εμπειρία που έχω, ερωτώ την Επιτροπή πώ κάνει την επιλογή, τα κονδύλια να τα αντλήσει από το Progress. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Γιατί το Progress είναι όχι το καταλληλότερο, εν περιπτώσει, κονδύλιο ή καταλληλότερη πηγή χρηματοδότηση Και ερωτώ γιατί. Διότι, από ό,τι φαίνεται, ενώ υπάρχει το το Jasmine, γιατί να χρησιμοποιείτε αυτό ή δεν προτείνετε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά της ε, χρήσης του πρόγραμματος ως πηγής χρηματοδότησης ή υπέρ της δημιουργίας μιας ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό. Γιατί αυτή θα έχει το πλεονέκτημα ότι η δεν προτεινετε κατι διαφορετικο υπαρχουν πολλα επιχειρηματα κατα της χρησης του προγραμμα ως Επιτροπή θα είναι σε θέση να ελέγχει προκαταβολικά, χάρη σε αυτήν την ειδική γραμμή, τα ποσά τα οποία διαφορετικά θα άφηνε να ε, ελέγξουν και να κρίνουν αυτόνομα τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι η επιλογή του Progress δείχνει ότι δεν έχει γίνει σωστά η δουλειά, απλώς και μόνο. Δεν έχει γίνει αρκετά προσεκτικά η επεξεργασία της πρότασης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική γραμμή, μια γραμμή πιλωτική ενδεχομένως με την ε, δοκιμαστική, αν θέλετε, εφαρμογή των ε, ε, μικροπιστώσεων και στη συνέχεια να πούμε έχουμε το Jasmine που ε, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αναλάβουν τη δράση αυτή με βάση την εμπειρία που έχουμε από, τις δοκιμαστικές, ε, από τη δοκιμαστική περίοδο και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Το progress το ίδιο είναι μία βάση η οποία αφορά Ε, ομάδες οι οποίες δεν θα είχαν καμία δυνατότητα για πίστοση που ε, και σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την δικτύωση. γιατί δικτύωση δεν χρειάζονται πιστώσεις, δεν χρειάζονται κονδύλια και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η επιλογή του Progress. Ρωτώ λοιπόν την εισηγήτρια εάν, δεδομένου ότι η κυρία Χάρκιν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην υπόθεση αυτή, ε, θα ήταν σκόπιμο να την συμβουλευθεί για να ακούσει τι ιδέες θα μπορούσε να ε, προτείνει και να φροντίσουμε στη δική μας πρόταση να αποφύγουμε την, ε, ε, το να τεθούν στο περιθώριο ορισμένες ομάδες που φαίνεται ότι ε, αποκλείονται αυτομάτως. Εσείς μιλήσατε για τους Ρωμά, επί παραδείγματι. Από την ε, πρόταση της Επιτροπής φαίνεται ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση. Γιατί λοιπόν ε, να μην δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ε, την, ε, κάποιες ομάδες συγκεκριμένες ε, πολιτών κατά τρόπον ώστε να επιτρέψουμε στο πρόγραμμα να προχωρήσει έτσι πειραματικά και ταυτόχρονα με μια ειδική γραμμή στον προπολογισμό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και να πω ότι το θέμα των μικροχρηματοδοτήσεων και μικροπιστώσεων έχει ιδιαίτερη έγκλη γιατί εδώ και χρόνια δίναμε τον αγώνα μας παρασκηνιακά για ορισμένες πρακτικές ε, χωρών όπω η Ουγγαρία και σήμερα ξαφνικά το θέμα αυτό έχει γίνει το απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε συζήτηση για τη διέξοδο από την κρίση. Και το γεγονό ότι ακόμη και η G20 ανέφεραν αυτό το θέμα δείχνει πόση σημασία έχει αποκτήσει το θέμα των μικροχρηματοδοτήσεων. Και υπάρχει βέβαια αυτός ε, ο ενθουσιασμός, ο προφορικός, αλλά δεν θα πρέπει να χαθούμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τα έργα. Γιατί η έμπρακτη εφαρμογή των προτάσεών μας είναι το ζητούμενο εδώ. Θα πρέπει καταρχήν να εντοπίσουμε περί τίνος πρόκειται και να το οριοθετήσουμε. Γιατί στον τομέα αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος σύγχυσης. Αν εγκαινιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία που υποστηρίζαμε εδώ και χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στόχος μας είναι να καλύψουμε μια ιδιαίτερη ανάγκη που υπάρχει. Και η ανάγκη αυτή δεν θα είναι εναλλακτική ε, ρύθμιση σχέση με τα αισθήματα κοινωνικής προστασίας, ούτε θα είναι μία προέκταση των ε, προβλημάτων χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι μια πρακτική ενδιάμεση που έχει ιδιότυπο χαρακτήρα και που προσπαθεί να καλύψει ταυτόχρονα και οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε όμως ένα τέτοιο πρωτότυπο τρόπο χρηματοδότησης για να επαναφέρουμε στην αγορά εργασίας άνθρωπους που δεν θα ήταν με διαφορετικό τρόπο. Απλώς θέλουμε να δώσουμε σε ορισμένους την ευκαιρία να καταφέρουν μόνοι τους ουσιαστικά να επανέλθουν στην αγορά απασχόλησης. Οπότε διαρωτώ με κατά πόσο είναι σκόπιμο να καλύψουμε στην ίδια πρόταση και τα θέματα της αποταμίευσης και διάφορες ε, δομές αποταμίευσης, γιατί αυτές υπακούν σε διαφορετική λογική. Σε πολλές χώρες βέβαια είχαμε κάποια credit unions που ήταν χρήσιμες δομές ε, έκφρασης αλληλεγγύης και κινητοποίησης γιατί πραγματικά βρίσκονται κοντά στους ε, έχοντες ανάγκη, αλλά αν στις μικροπιστώσεις, στις μικροχρηματοδοτήσεις ε, συμπεριλάβουμε και την μικροαποταμίευση, πιστεύω ότι θα απομακρυνθούμε από τον πρωταρχικό μας στόχο. Κάτι που θα ήταν εσφαλμένο κατά τη γνώμη μου. Επίσης, πιστεύω ότι πίσω από ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είμαστε χαλαροί σε ό,τι αφορά τι συνθήκε πρόσβαση των δικαιούχων. Μιλούμε για ευάλωτε ομάδε που έχουν δύσκολα πρόσβαση σε κονδύλια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση εκτό από το οικονομικό σκέλος, στο σκέλο τη καθοδήγηση, τη κατάρτιση και τη παρακολούθηση τη εφαρμογή του προγράμματο. Και θα συνεννοηθώ με τους συντονιστές για τις ε, μελλοντικές μας πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ώστε να εξετάζουμε σε κάθε κράτος μέλος τι δομές υπάρχουν που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τέτοιων προτάσεων. Ώστε, όπως είπατε, να υπάρχει διαφάνεια και στην ανταλλαγή ε, πληροφοριών και πρακτικών και να δούμε πώς εφαρμόζονται εμπράκτως οι πρωτοβουλίε αυτές στα κράτη-μέλη. Ορισμένε κλασικές δομές χρηματοδότηση των επενδύσεων, συνεταιριστικέ ή τραπεζικές, δεν βλέπουν με καλό μάτι τέτοιου είδους ε, χρηματοδοτήσει, Έχοντα την αίσθηση ότι θα είναι ανταγωνιστικές με τη δική τους δραστηριότητα. Γιατί ξεχνούν ότι εμείς καλύπτουμε μία πρόσβαση σε πιστώσεις που οι οργανισμοί αυτοί δεν τις καλύπτουν. Πιστεύω ότι αν οργανώσουμε μια ημερίδα μελέτης με το θέμα αυτό θα ρίξουμε περισσότερο φως στο μηχανισμό αυτό για να διασκεδαστούν οι αμφιβολίες. Και η τελευταία μου παρατήρηση αφορά τη δημοσιονομική γραμμή. Η Επιτροπή μας ήδη έχει αποφαθεί για αυτό το θέμα. Όταν εκπονούσαμε την γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό 2010 με εισηγητή τον κύριο Ορή, είχαμε ψηφίσει υπέρ μιας αυτοτελούς δημοσιονομικής γραμμής για τις μικροχρηματοδοτήσεις γιατί ούτε το Progress ούτε το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, ήταν τα κατάλληλα ταμεία για να χρηματοδοτήσουν αυτό το νέο μέσο. Άλλωστε, τα κονδύλια των δύο προγραμμάτων έχουν ήδη προσημειωθεί. Δεν θα ήταν σωστό λοιπόν να απομυζήσουμε το πρόγραμμα Progress για να χρηματοδοτήσουμε τις μικροχρηματοδοτήσεις. Γιατί μπορεί κάτι τέτοιο να ικανοποιούσε το Συμβούλιο, αλλά εμείς δεν συμφωνούμε με μια τέτοια πρόταση. Και αυτό συμφωνώ απόλυτα με την πρότασή σας για μια ξεχωριστή αυτοτελή δημοσιονομική γραμμή για τη χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας και όχι από τα κονδύλια του Progress. Αυτό άλλωστε είχαμε ψηφίσει με τη γνωμοδότησή μας για τον προϋπολογισμό. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των ομιλητών, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την υποστήριξή του, έτσι τουλάχιστον εγώ το κατανόησα. Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία, αλλά υπάρχουν σημεία συμφωνίας τα οποία θα χαρακτήριζα χρήσιμα. Ευχαριστώ επίσης και για τα σχόλιά σας. Τα σχόλια σαφώς βελτιώνουν και ε, σε επίπεδο λεπτομέρειας διευκρινίζουν το κείμενο. Άκουσα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τις ε, προσδοκίες τις μεγάλες που υπάρχουν από ένα τέτοιο πρόγραμμα, από την πολύ μεγάλη ζήτηση που μπορεί να υπάρξει, είπατε ορισμένη, κάποιοι άλλοι ανησυχείτε από την μικρή ζήτηση η οποία αναμένεται να υπάρξει κάποια επιπλέον σχόλια. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι η συζήτηση που έγινε για το ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα, ποιοι μπορεί να είναι οι δικαιούχοι. Και υπήρξε και μάλιστα ε, μια απόψη η οποία λέει ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα κατάλογο πιθανών δικαιούχων, αλλά να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να εντοπίσουν διαφορετικού τύπου ομάδες που έχουν ανάγκη. Σε κάποιες χώρες οι νέοι σαν παράδειγμα μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Σε κάποιες άλλες χώρες απαιτείται περαιτέρω στήριξη για τους Ρώμα, για τους ηλικιωμένου, για τις γυναίκες κτλ. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να βρω μια διαφορετική ισορροπία Άκουσα με ενδιαφέρον επίσης ότι πολλοί πιστεύουν όπως και εγώ ότι το πρόγραμμα Progress δεν είναι η κατάλληλη τουλάχιστον δημοσιονομικά γραμμή και αυτό για πολλούς λόγους. Είπατε ότι εφόσον δεν απορροφηθεί επαρκώς το Progress τότε είναι δική μας ευθύνη αυτοί οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Progress αλλά δεν είναι σε θέση να ωφεληθούν από αυτό να έχουν μια διαφορετική ευκαιρία. Αυτό βέβαια δεν είναι λόγος για να μειώσουμε τις πιστώσεις τις οποίες έχει το πρόγραμμα στη διάθεσή του. Το θέμα δεν είναι να κρίνουμε αν τα χρήματα αυτά είναι ε, θα έλεγα αντίστοιχα του ύψους των πιστώσεων που έχουμε διαθέσιμες για το πρόγραμμα σαν παράδειγμα αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης Τα παρουσιάζω λίγο συνθετικά αυτά που έχω να πω. Το θέμα είναι και σε ποιο βαθμό μπορούμε να εμπλέξουμε τα εμπορικά πιστοτικά ιδρύματα. Αν το κάνουμε αυτό θα σημειώσουμε ένα σημαντικό βήμα. Εφόσον οι πιστωτικές, αυτές, ε, οι πιστωτικές, τα πιστοτικά αυτά ιδρύματα, οι τράπεζες, εν πάση περιπτώσει αυτές, θεωρήσουν ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή μπορούν να αγκιστρώσουν περισσότερους πελάτες, τότε Πράγματι αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για μας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι δεν θα θεωρήσουν ότι οι εμπορικές τράπεζες αντιμετωπίζουν κινδύνους μέσω της συμμετοχής τους από το πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Σύντομα, να πω κάτι στο οποίο αναφερθήκατε εσείς, ότι είναι πολύ περίπλοκα γραφειοκρατικά τα ταμεία αυτά. Νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες γίνονται εδώ είναι μια εγγύηση ε, έτσι ώστε οι διαδικασίες να παραμείνουν σχετικά απλές. Το θέμα είναι να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό για την σωστή κατάρτιση των πιθανών δικαιούχων και τη σωστή τους ενημέρωση έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Το θέμα δεν είναι η εναρμόνιση μόνο των κοινοτικών μέτρων και των εθνικών, αλλά και σε επίπεδο οργανωτικό να καταλήξουμε σε μια διαδικασία η οποία να είναι κατανοητή. Προφανώς ένα επίπεδο εναρμόνισης απαιτείται. Λοιπόν, κλείνοντα λίγο, μου ζητάτε να τελειώσω. Προφανώς δεν πρόκειται για πανάκια η συγκεκριμένη πρόταση. Είναι ένα από τα μέσα τα οποία μπορούν να καλύψουν μια ανάγκη η οποία υπάρχει, μια πραγματική ανάγκη, και νομίζω ότι θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο το Ταμείο αυτό. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Επ' αυτή τη βάσεως και επ' αυτή τη συγκεκριμένη ανταλλαγής που προηγήθηκε θα ορίσουμε την επόμενη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών την 6η Οκτωβρίου 18η απογευματινή και θα ψηφίσουμε την 5η Νοεμβρίου σύμφωνα πάντα και με το ημερολόγιο σε εισαγωγικά που θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπε επιτροπές. Λοιπόν, υποδέχομαι εδώ τον κύριο Σπίτλα για την πρώτη ακρόαση από την αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου. Θα του δώσω το λόγο αμέσως. Θα ήθελα όμως να ζητήσω από όλους τους ορθίους στην αίθουσα να πάνε στη διπλανή αίθουσα, στην αίθουσα ακρόασης και να σταματήσουν τις κατηδίαν συζητήσεις διότι μας ενοχλούν. Το λέω και στην Αγγλική λέει η Πρόεδρος και λέει το ίδιο πράγμα. Personal conversation. It's just not possible to have this noise in the room while people are, are, are speaking. Thank you for your understanding. Monsieur le Commissaire, merci. Λοιπόν κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη θα έλεγα φάση σε σχέση με το δικό σας χαρτοφυλάκιο η κατάσταση στην απασχόληση παραμένει ασταθής, οι δείκτες μπορεί να οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα, αλλά η απασχόληση εξακολουθεί να υποφέρει. Γι' αυτό λοιπόν η δική σας φωνή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε κάποια νομοθετικά μέσα μπροστά μας, τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Αυτές τις συζητήσεις προσπαθούμε να εμβαθύνουμε για να παρακολουθήσουμε σωστά την πολιτική την οποία ακολουθείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό η συνεισφορά σας θα είναι πολύτιμη. Σας ζητώ όμως να είστε σύντομος έτσι ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν και να σας ακούσουν αλλά και να κάνουν αυτό που πάντα προτιμούν, δηλαδή να σας θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερω που βρίσκομαι ενώπιον σα σήμερα. Ευχαριστώ κυρίω πρώτα απ' όλα την κυρία Μπέρε που μου δίνει την ευκαιρία να εκφραστώ ενώπιον σας και θα ήθελα ιδιαίτερα να σας συγχαρώ για την πρόσφατη εκλογή σας ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφέ ότι η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι διαφορετική από αυτήν που είχαμε στο παρελθόν. Το 2004 το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίαζε μια ανάπτυξη 22,5% και το 2009 κατά τις εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μειωνόταν κατά 4%. Όσον δε αφορά την ανεργία. Το Μάιο του 2004 είχα μια είχαμε μια διαρκή πτώση μέχρι το 2008 πέφτω στο 7%. Το 2009 όμως τον Ιούλιο ήταν 9,2% του ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και να φτάσει μέχρι το 11,5% το 2010. Επίσης θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τις κοινωνικές ανησυχίες προκαλεί η κρίση που υπογράμμισαν και οι Υπουργοί Απασχόλησης του όσα σε συνεδρία στην οποία έλαβα και εγώ μέρος ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει πραγματική διέξοδος από την κρίση όσο δεν έχει σταθεροποιηθεί η απασχόληση. Όσο δηλαδή δεν έχουμε ε, θετικό ισοζύγιο δημιουργίας της συνεργασίας. Κυρίε και κύριοι, η κρίση που διανύουμε είναι η σοβαρότερη από το πέρας του, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είπε και εκθέτοντας τις πολιτικές του κατευθύνσεις για την προσοχή εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Παρόσο, έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Έχουμε να κάνουμε κυρίως και επιπλέον με μια κρίση αξιών πάνω στις οποίες είναι χτισμένη και θεμελιωμένη η οικονομία μας, η κοινωνία μας. Όσο τραγική λοιπόν να είναι αυτή η κρίση, δεν πάβει να αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία, πραγματική ευκαιρία, σε κάθε επίπεδο και όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κοινωνία στηρισμένη την ε, στη γνώση και με χαμηλό ε, ίχνος άνθρακα και επίσης μια κοινωνία που θα μπορεί κανείς να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. Τα τελευταία 100 χρόνια ο μιλητή δυστυχώς δεν χρησιμοποιεί τη μετρική του γλώσσα και είναι δυσνόητος τουλάχιστον. Είχαμε πολύ σοβαρές κρίσεις και θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα, λέει ο μιλητή. Ανεπτύχθη εταιρική σχέση για την αναδιάρθρωση μέσα από φόρουμ αναδιάρθρωσης. Και όταν γίνεται αναπόφευκτη μια αναδιάρθρωση, πρέπει να προσφέρεται υποστήριξη στους ε, απολυθέντες. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης το 2007 και το αναθεωρεί το 2009, το οποίο από τη σύστασή του έχει προσφέρει υποστήριξη σε 26.000 εργαζομένους και από την αρχή του έτους έχει λάβει πολλές, πολλά νέα αιτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι χάρη και στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να, τα, να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά το χειρότερο δυνατό. Ενισχύουμε επίσης το ρόλο του, της Επιτροπής Επιχειρήσεως και ιδιαιτέρως χαίρομαι για την πρόταση μας του 2008 που υιοθετήθηκε πολύ γρήγορα χάρη στην, Ευρωπαϊκή, στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης ε, προβάλαμε, προάγαμε τον κοινωνικό διάλογο με ιδιαίτερη έμφαση στον εργαζόμενο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υιοθετήθηκαν αυτόνομες συμβάσεις και συμφωνίες ε, για την καταπολέμηση του στρες και των προβλημάτων ψυχολογικού χαρακτήρα στη χώρα εργασία και άλλα ζητήματα τα οποία λαμβάνουν πλέον τη μορφή της ε, οδηγίας όπως η γονική άδεια και η ε, αποτροπή τραυματισμών από οξέα αντικείμενα. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με την βελτίωση των δεξιοτήτων και με την ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2008 για τις νέες δεξιότητες, για νέες θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων έως το 2020 για καλύτερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, ανταποκρινόμενα στην κρίση τα κράτη-μέλη υιοθετούν σχέδια ανάκαμψης που επιβαρύνουν βαρύτατα τους εθνικούς προϋπολογισμούς, σχέδια ανάκαμψης που εν όλο επέτρεψαν την αποτροπή των αρνητικότερων επιπτώσεων της κρίσης. Οι ρήτρε κοινωνικής προστασίας έχουν μπορέσει να σταθεροποιήσουν την κοινωνική κατάσταση, πριν όμως τα σχέδια ανάκαμψης έχουν και το τίμημά τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω της κρίσης οι δαπάνες ε, κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει από το 20% επί του ΑΕΠ το 2008 στο 31% το 2010. Ταυτόχρονα τα έσοδα των κρατών μελών αναμένεται ότι θα μειωθούν σημαντικά λόγω της, ε, του περιορισμού της, της περιστολής των δραστηριοτήτων. Η κρίση επίσης καθιστά ακόμη πιο επίγουσα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μακροπρόθεσμα όπως οι αλλαγές στη δημογραφική ε, κατάσταση στην Ευρώπη. Έχουμε ένα περιθώριο ευκαιρίας, θα έλεγα, δεκαετίας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας γυράφουσας κοινωνίας. Το 2005 προτείναμε μια πράσινη βίβλο για τις δημογραφικές αλλαγές. Και εγώ προσωπικώς υπέβαλα και νέες προτάσεις πρωτοβουλίας για την προαγωγή της, ε, του συνδυασμού του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου ε, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άδεια μητρότητας και την ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν αυτοί έχουν ανεξάρτητη δραστηριότητα και επίσης ε, πέρυσι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σχέδιο οδηγίας για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην γονική άδεια με το σύστημα του ανοιχτού συντονισμού στην κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση έχουμε προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών γύρω από κοινού στόχους και προσπαθούμε να ε, εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με όρους όμως και ισότιμους, ισότιμης κατανομής μεταξύ των γενεών και βιωσιμότητας ως ε, νέος επίτροπος από νέο κρατος μέλος είχα ως καθήκον να ε, ρίξω τα όρια και τους φραγμούς μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών παρά τα μεταβατικά μέτρα ε, απαγόρευσης ρεύθυνσης κυκλοφορίας των εργαζομένων από τα νέα κράτη-μέλη και με χαρά και ικανοποίηση διαπιστώνω ότι πέντε χρόνια μετά την ένταξη του 2004 η οι πήκοοι των νέων κρατών μελών έχουν δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας 13 από τα 15 ε, παλαιά κράτη-μέλη. Οι δε Βούλγαροι και Ρουμάνοι εργαζόμενοι μπορούν ελεύθερα να εργαστούν σε 15 από τα 25 προηγούμενα μέλη. Για μένα η διεύρυνση αποδεικνύεται έτσι ως επιτυχής. Και βεβαίως για μένα το να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά εργασίας δεν ισοδυναμεί με τη δημιουργία μιας ε, άνομης αγοράς εργασίας, χωρίς κανόνες δηλαδή. Και έτσι πιστεύω ότι με πολύ, ότι με πολύ μεγάλη επιτυχία η θέσπιση του κανονισμού 493 για την εφαρμογή του συστήματος κοινωνικής προστασίας Επίσης έχουμε μεριμνήσει για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο πολύ, ένα ζήτημα για το οποίο επαναλημμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Κατά την ακρόαση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου θα ακούσατε τον πρόεδρο Μπαρόσο που δεσμεύτηκε να ε, υποβάλει νέα πρόταση σχετικά, σχετική με την θέση σε εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης, προσφέρουμε προστασία και για τη βελτίωση, μάλλον προσφέρουμε, δίνουμε την προτεραιότητα στην βελτίωση προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων και με χαρά βλέπω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπόρεσαν εν τέλει να καταλήξουν συμφωνία Ω προ την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποσκοπεί στην ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων interim σε συμβόλαιο, δηλαδή μικρή διάρκεια. Λυπούμε που δεν μπορέσει να συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο ω προ την αναθεώρηση τη οδηγία για το χρόνο εργασία, όπω γνωρίζετε ο Πρόεδρος Παρόσο δεσμεύθηκε στην υποβολή νέα πρόταση μέχρι το καλοκαίρι του 2010 αφού γίνει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εις βάθος ανάλυση της κατάστασης και η Επιτροπή θα αναζητήσει ε, ισότιμες και βιώσιμες λύσεις ε, που δεν θα οδηγήσουν σε οπισθοδρόμησης προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνίστηκα με πάθος ε, προσπιζόμενος το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Σημειώσαμε κάποιε ήττε, αλλά πάνω απ' όλα νίκε. Και πάντω, δεν μπορούμε να επαναπαυόμεθα στις δάφνες μας και θα πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγική διεξόδου από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Νοέμβριο του 2008 αντέδρασε αποφασιστικά ε, ενώψη ε, ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης και τον Ιούνιο του 2009 υιοθέτησε ανακοίνωση με τίτλο ε, κοινή δέσμευση, κοινή στράτευση για την απασχόληση με τρεις κύριες προτεραιότητες στο πρόγραμμά μας, δηλαδή διατήρηση στο χώρο, στην θέση εργασίας του εργαζομένου, προαγωγή της κινητικότητας, βελτίωση της εργασίας, δεύτερον βελτίωση των δεξιοτήτων και καλύτερη ανταπόκριση ανάγκες της αγοράς εργασίας και τρίτον προαγωγή ε, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και επίσης υποστηρίζουμε και τις προσπάθειες των κρατών μελών προτείνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απλούστευση των ε, κανόνων ε, λειτουργίας του ε, κοινωνικού Ταμείου, διευκόλυνση των κρατών μελών και 100% χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη σε σχέδια που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2009 και 2010. Αυτή ήταν η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δυστυχώ αντιμετωπίζει αντίσταση από πολλά κράτη-μέλη. Και όπως είπα και νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσαρμόσει τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση της, το καλύτερα να ανταποκριθεί στους, ε, στα δεδομένα της τωρινής κρίσης. Προηγουμένως είχε μία πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση ενός νέου μέσου για τις μικροπιστώσεις, την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Ένα θέμα το οποίο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την συγκεκριά σας κυρία Αγκούνς και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καταλήξουν σύντομα σε συμβαστική λύση. Η τρέχουσα κρίση, όπως είπα, αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των κοινωνιών μας και έτσι η στρατηγική για τη διέξοδο από την κρίση θα πρέπει να συνδυαστεί με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ιδίως δηλαδή και επί παραδείγματι διαχείριση της μετάβασης ή των της σε ε, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με θετική με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη, με ανεπτυγμένη την, ε, ανεπτυγμένα τα ποσοστά των, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020, που σημαίνουν ταυτόχρονα και περισσότερες θέσεις εργασίας, περίπου τα 400.000 και 0,24 ε, ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ανάπτυξη μιας νέας ατζέντα για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής Λισαβόνας, αλλά και μετά Λισαβόνα στις ε, σχετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, καταθέσει στις αρχές του προσεχούς έτους. Είναι όμως πιστεύω σαφές ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής Λισαβόνας ιδιαίτερου προκειμένου να ληφθεί υπόψη οι κατάσταση που αντιμετωπίσουν οι πιο ευάλωτε συμπολίτε μα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι δημογραφικέ αλλαγέ εν των οποίων πρέπει να αναθεωρηθεί το συνταξιδοτικό σύστημα και το σύστημα γιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή θα είναι οι κύριοι τομεί στου οποίου θα πρέπει να, ε, να σκύψουμε, όπως επίσης και στη μεταναστευτική πολιτική. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε το ζήτημα της αγύρανσης των κοινωνιών μας, να προλάβουμε τις εξελίξεις και ιδιαίτερα αναφέρομαι στην νομοθεσία κατά των διακρίσεων, διεθνή νομοθεσία. Επίσης σκέφτομαι, στη, έχω υπόψη μου τις ε, Διεθνή Συμβάση των Εθνών υπέρ των ατόμων με αναπηρίες και τη απασχόλησή τους ή της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρώμα. Κυρίες και κύριοι, η κρίση των δείχνει ότι οι βάσεις του κοινωνικού μας μοντέλου είναι γερές. Τα κράτη-μέλη αντιδρούν με τρόπο αποφασιστικό και τώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας για να διαφύγουμε από την κρίση και να αναπτύξουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η βάση συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ γερή και θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα προσεχή έτη κατά την απόψή μου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που σας ανέφερα. Και για να τελειώσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία τις τελευταία, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταια αυτά πέντε χρόνια και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την επόμενη πενταετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. <coughs> Οι βουλευτές σας άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά ζήτησαν 19 το λόγο με πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα υποβάλουν ερωτήσεις. Όλοι θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Οπότε δεν θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε στις 5, αλλά στις 5 και 4, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα δίλεπτο στον καθένα για να θέσει τις ερωτήσεις του. Πρώτα η κυρία Λίν, μετά ο κύριος Φάλμπρ. Θα ακούμε ένα τρεις τους ομιλητές και μετά μέσα σε ένα πεντάλεπτο θα πρέπει να απαντάτε. Περιορίζω και το δικό σας χρόνο δηλαδή απαντήσεων. Κύριε Ελλήν, πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και πάλι τον Επίτροπο για το έργο του για την καταπολέμηση των διακρίσεων την τελευταία πενταετία. Ελπίζω να παραμείνετε στη θέση σας για να συνεχίσετε το αξιέπαινο έργο που έχετε ξεκινήσει στον τομέα αυτό. Μήπως ξέρετε πότε το Συμβούλιο θα κάνει κάτι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, έχουν δράσει. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι, δεν κάνω λάθος, έχουν καταλήξει συμφωνία. Πότε θα υποβληθεί πρόταση για, τις, για τους τραυματισμούς από βελόνε ε, σύριγγων. Γιατί νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους τραυματισμούς από βελόνε. Αναφερθήκατε και στο θέμα της γύρας του πληθυσμού. Προβλέπετε να γίνει κάποιο έργο, να αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία για, τις, για πιο μακροπρόθεσμη παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, γιατί έχουν γίνει πολλές έρευνες στο θέμα αυτό, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε ένα δεντολογικό κώδικα για τέτοια μακροπρόθεσμη φροντίδα σε ηλικιωμένους ή να συνάψουμε μια ευρωπαϊκή συνθήκη για τους ηλικιωμένους ε, κατ' εικόνα και ομοίωση της ε, συνθήκης ε, για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτά είναι τα βασικά μου ερωτήματα. Ο κύριος Φάρμπλ και μετά η κυρία Πασκάλ Γκρούνη. Συχνά, α, ακούγοντας τον Επίτροπο, ε, σκεφτόμουν ότι φαίνεται σαν ο πλανήτης ζούσε την τελευταία πενταετία. Γιατί είδαμε ότι το κοινωνικό μας μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε πολλές επιθέσεις, η επιρροή των συνδικάτων αποδυναμώνονταν, ε, ε, ο κοινωνικός διάλογος ήταν φαρσοκομωδία σε πολλές χώρες, ε, η στρατηγική της Λισαβόνας έχει γίνει περίγελος και κανένας δεν τη σέβεται και η οδηγία για την, για την εργασία, για το ωράριο εργασίας, η οδηγία για τις υπηρεσίες, όλα αυτά δεν προχώρησαν. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένο ούτε από το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινωνικά θέματα, αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένο ούτε και από το προσωπικό έργο του Επιτρόπου στον τομέα αυτό. Έχω μία ερώτηση για να μην τρώω χρόνο και από τους συναδέλφους. Εκπονείται ε, η σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας και τα συνδικάτα διαμαρτύρονται γιατί στην Κορέα καταστρατηγούνται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η Κορέα δεν έχει εγκρίνει σχεδόν καμία από τις συμβάσεις και συμφωνίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη και η θέση του Επιτρόπου για την προετοιμασία της σύναψης συμφωνίας με την Κορέα. Η κυρία Γκρούνη έφυγε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Μάν. Ähm, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, οπότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ευέλικτη ασφάλεια, flex security. Και είπατε θα πρέπει να γίνει η ανάλυση της κατάστασης ορισμένα κράτη-μέλη για τις ανάγκες σε επενδύσεις. Πώ θα το κάνετε αυτό. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δεξιότητες, αλλά πώ θα γίνει αυτό. Θα κάνουμε την ανάλυση μας όποτε έχουμε χρήματα ή θα έχουμε μια πιο ε, διαρκή ε, διαδικασία. Κάτι ακόμη. Εμένα στην εκλογική μου περιφέρεια ξέρω ότι υπάρχει η επιχείρηση της Opel. Έχουμε λοιπόν προβλήματα ε, σε σχέση με το κλείσιμο των μονάδων παραγωγής και ο μόνος με τον οποίο έχουμε να κάνουμε ε, είναι η Επίτροπος η αρμόδια για τον ανταγωνισμό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το κρατήδιο της ΕΣΥ στο οποίο βρίσκομαι εγώ, ε, αλλά και για τις κάτω χώρες και για άλλες εγκαταστάσεις οι μονάδες της Όπελ. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Επίτροπος ο αρμόδιος για τα κοινωνικά θέματα και την προστασία των εργαζομένων που απολύονται είναι όλα αυτά συμβατά σε τελευταία ανάλυση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα ελέγχετε ή μήπως τα αφήνετε στα χέρια του ή καλύτερα τη συναδέλφου που ασχολείται με τον ανταγωνισμό. Κύριε Επίτροπε, αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε. Πολύ ευχαρίστω. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί και η Σουηδική Προεδρία έθεσε το θέμα αυτό επιτάπητο στο Συμβούλιο. Οπότε αναμένεται πρόοδος αλλά με αργό ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα. Μετά από πολύ χρόνο καταλήξαμε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, καταλήξαμε σε ένα ε, μεστό και τεκμηριωμένο κείμενο που θα μετατραπεί σε οδηγία. Και νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο στο θέμα της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Σε ό,τι αφορά τη δημογραφία, τα δημογραφικά προβλήματα και την ε, ποιοτική φροντίδα. Σίγουρα οι δημογραφικές αλλαγές έχουν αποφασιστική σημασία. Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά σε πολλά συστήματα εθνικά υπάρχουν κενά και αδυναμίες. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αδυναμία εντοπίζεται στην παροχή μακροχρόνιας φροντίδας. Γιατί εκεί δεν έχουμε εξεζητημένες στρατηγικές στα κράτη-μέλη. Έχουμε προκαλέσει μια συζήτηση για το θέμα αυτό, μια συζήτηση που θα έχει τεράστια σημασία και που ευελπιστούμε ότι θα καταλήξει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τις χώρες μέλη, ενός θεσμικού πλαισίου που και ο θελός θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσει του κυρίου Ρίχαρτ Φάλμπρ, που είναι και συμπατριώτης μου και μάλιστα ε, τέλεσε και γερουσιαστή στην Τσεχία. Είναι παλιός γνώριμος λοιπόν. Θα ήθελα να του πω λοιπόν ότι όλα αυτά που σας ανέφερα στην ε, ομιλία μου δεν είναι καθόλου ουτοπικά και εξωπραγματικά. Αποτελούν πραγματικότητα, αθιαφισβήτητη πραγματικότητα. Και είναι αλήθεια ότι Μερικές ε, επιχειρήσεις πάγωσαν για πολλά χρόνια, για μία οκταετία, αλλά νομίζω ότι βελτιώσαμε την ποιότητα του έργου των ε, εργασιακών συμβουλίων και τα αποτελέσματα φάνηκαν και στην περίπτωση της Όπελ. Οπότε αν έχουμε κάποιο όραμα και δεν έχουμε αρκετή οξυδέρκεια, μπορεί όντως η αντίληψη της πραγματικότητας που θα διαμορφώσουμε να είναι εσφαλμένη. Πάντως, δεν συμφωνώ με την διαπίστωσή σας ότι η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε. Αυτή είναι η δική σας υποκειμενική και μεροληπτική γνώμη. Γιατί μπορεί μεν η στρατηγική της Λισαβόνας να μην υλοποιήσει όλους τους στόχους, αλλά σίγουρα ορισμένους τους εκπλήρωσε, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα. Εκεί βλέπουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει πολλούς στόχους μας. Σίγουρα έχει κενά και η στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά τίποτα δεν είναι τέλειο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την απαρνηθούμε και να μην την εφαρμόζουμε. Άλλωστε, τη στρατηγική της Λισαβόνας τη μιμήθηκαν σχεδόν κατά γράμμα και οι Ιάπωνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται υπόδειγμα η στρατηγική αυτή σε πολλά σημεία του πλανήτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, σύναψη συμφωνίας με την Κορέα, πιστεύω εν γέννη ότι η διαμόρφωση ενός χώρου ελεύθερων ε, συναλλαγών και η δημιουργία ενός δίκαιου εμπορικού χώρου και θεμητού είναι αξιέπαινο στόχος. Και αυτό είναι ο στόχος που επιδιώκουμε σε όλες μας τις εμπορικές συμφωνίες. Για τη συνθήκη της Κορέας συγκεκριμένα, έχω αποστείλει επιστολή κρούντας τον κόδωνα του κινδύνου για μια πιο προσεκτική και αργή πρόοδο. Στην επιστολή αυτή εξέφρασα πολλές ε, ε, αμφιβολίες και δισταγμούς και είπα ότι ίσως είναι σπευσμένο να προβούμε σε μια ταχεία σύναψη αυτής της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Όπελ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ως συλλογικό όργανο, αφενός αφετέρου όμως υπάρχει ένας επιμερισμός των ευθυνών και των καθηκόντων. Το θέμα της αναδιάρθρωσης της Όπελ και η σχέση της με την εσωτερική αγορά είναι αρμοδιότητα της συναδέλφου Νέλη Κρούς και όχι δική μου. Μόνο τα κοινωνικά ζητήματα που απορρέουν από την υπόθεση Όπελ είναι δική μου αρμοδιότητα. Ή τα θέματα ενημέρωσης των εργαζομένων. Όλα αυτά τα θέματα τα έλεγξα και διαπιστώνω τις όλες οι οδηγίες που αφορούν την διαβούλευση και την ενημέρωση των εργαζομένων έχουν γίνει σεβαστές στην περίπτωση της Όπελ. Και το Εργασιακό Συμβούλιο της Όπελ είναι ιδιαίτερα δραστήριο και προσπαθεί να διεκδικήσει μια ευρωπαϊκή λύση. Και πέραν της ε, πιθανότητας χρήση των κονδυλίων του ΕΚΤ για την ε, αναδιάρθρωση της Όπελ, και εκεί ήμουν σαφής ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν την παρακολούθηση, τη στήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών και τον σεβασμό των διατάξεων για τα εργασιακά συμβούλια. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε τις φαιές και θολές ζώνες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά όμως τα λάβαμε υπόψη και εξακριβώσαμε τη συμβατότητά τους ε, με τους εμπορικούς με τους ε, κοινοτικούς κανόνες. Παρακολούθησε τις διαπραγματεύσεις από την αρχή και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει όλες αυτές τις αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Η κυρία Σόιτερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας αποκαλύψετε ένα τουλάχιστον μυστικό. Ξέρετε ότι αυτά που ακούσαμε στην Ολομέλεια σχετικά με την οδηγία για τις αποσπάσεις ήταν λίγο περίπλοκα. Ο κ. Μπαρόσο μας είπε ουσιαστικά, ο Προεδρός σας, ότι δεν θα τροποποιηθεί η συγκεκριμένη οδηγία για τις αποσπάσεις, αλλά θα δημιουργηθεί αντίθετα ένας κανονισμός, ο οποίος θα διασφαλίζει την ισότητα αμοιβή για την ίση εργασία. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν γύρω από τη συγκεκριμένη υπόσχεση του κυρίου Μπαρός. Και πώς ένας κανονισμός μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, ενώ γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την συμβατότητα ανάμεσα στα διαφορετικά κοινωνικά συστήματα που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε εγγυήσει για την επιτυχή εφαρμογή και σεβασμό του κανονισμού αυτού στις διάφορες χώρες. Πείστε μας για το αντίθετο αν πιστεύετε κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Για το 100% και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα αποσύρει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εμένει στην πρόταση. Και τι θα γίνει επίσης με το πακέτο του κανονισμού για την οικονομική συγκυρία. Θα μας κάνετε κάποιες νέες προτάσεις, θα εμείνετε στις παλαιότερες. Και έτσι είμαι. Και μετά η κυρία Μπλινκεβιτσίουτε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Σπίτλα, λέει η κυρία Τσίμα. Υποθέτω ότι δεν ήρθατε εδώ ελπίζοντας ότι μετά από πέντε χρόνια δουλειά σας θα σας ε, προσφέρουμε μια μεγάλη ανθοδέσμη συγχαίροντάς σας ε, για τον απολογισμό της δουλειάς σας και τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απασχόλησης. Αποκλείεται. Ο απολογισμός σας είναι, θα έλεγα, σαφέστατα αρνητικός και, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα ισχνός. δεν έχετε προχωρήσει στις διορθώσεις τις οποίες είχατε καταλήξει σε σχέση με ε, τις πρώτες προτάσεις σας, οι οποίες δεν απέδωσαν και οδηγούμε σε μία ερώτηση. Η διάδοχή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα ζητήσουν, θα ζητήσουν μία αλλαγή στις κατευθυντήριες οικονομικές γραμμές και προς ποια κατεύθυνση. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η σχέση ανάμεσα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε εγγυήσει για θέσεις εργασίας αξιοπρεπής είναι ένα ζητούμενο και με ποιο βαθμό θα μπορέσετε εσείς να βοηθήσετε με τα μέτρα που θα πάρετε για να καταπολεμήσουμε την ένδυα η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν τα μέσα που τους χρειάζονται για να καταπολεμήσουν την φτώχεια. Γνωρίζετε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα για να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες για τους αστέγους Ξέρετε επίσης ε, το πρόβλημα που υπάρχει σε άλλες χώρες για τα άστεγα παιδιά που ζουν στους δρόμους. Ποια είναι η πολιτική σας γραμμή. Οι θέσεις τις οποίες εξέφρασε ο κύριος Μπαρόσο δεν μας λέγουν τίποτα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν αναλαμβάνεται καμία μα καμία ευθύνη. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίμα. Η κυρία Μπλικεβιτσίουτε. Και μετά ο κύριος Χέλμερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις ε, ευρωπαϊκές χώρες σε διαφορετικό βαθμό. Η Λιθουανία, όπως και κάποιες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ εκείνων όπου κατέρευσε περισσότερο το ΑΕΠ και αυξήθηκε ραγδαία η, η ανεργία μαζί ταυτόχρονα με την μείωση των κοινωνικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κοινωνική προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει κάποια εργαλεία για την αντιμετώπιση τη κρίση. Σκοπεύει λοιπόν να αλλάξει τους τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο περί προσωρινής ε, απαγόρευσης της ε, εθνικής συγχρηματοδότησης με εισαγωγή νέων κανόνων και με απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Χέλμερ. Και μετά μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε να μας δείτε. Με χαρά άκουσα ότι έχει μπορέσει να βοηθήσει ήδη 26.000 άτομα το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή 0,005% επί του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε λαμπρά. Επίσης, με χαρά ακούω ότι μπορείτε από ό,τι φαίνεται μέσα σε 10 χρόνια να κάνετε ε, διαρθρωτικές αλλαγές για τη δημογραφική ορολογιακή βόμβα. Σας υπενθυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια είχαμε την ε, εισαγωγή της, συνθήκης, ε, του προγράμματος Λισαβόνος μέσα σε δύο χρόνια, μέσα σε δέκα χρόνια θα είχε μετατρέψει την Ευρώπη στην πιο ανταγωνιστική κοινωνία του κόσμου και τώρα παραδέχεται δέκα χρόνια μετά εσείς ο ίδιος ότι είχε γίνει λιγότερο ανταγωνιστική και έχει μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και χαίρομαι επίσης που λέτε ότι το, παγκοσμι... το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, μπορεί να βοηθήσει τους ε, εργαζομένους, της... τους απολυθέντες μάλλον της εταιρεία Dell στην Ιρλανδία. Θα ήθελα πολύ συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για το θέμα αυτό, γιατί σκοπεύω να τις δημοσιοποιήσω και να τις δημοσιεύσω στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, διότι ερωτώ πώς είναι δυνατόν να τολμάτε να κάνετε χρήση κοινοτικών κονδυλίων για προεκλογικούς σκοπούς σε ένα κράτος μέλος στο, πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας. Ντροπή σας. Και επίσης, όπως είπε και η πρόεδρος τελευταία ανάλυση, υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, αν θέλετε να την το, να θέσετε σε λειτουργία το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, πρέπει να έρθετε στο Κοινοβούλιο και να στήσετε την αδειά του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, από ό,τι φαίνεται, έκανε την ανακοίνωσή του χωρίς καν να ερωτήσει το Κοινοβούλιο. Επειδή ότι μιλούμε για δημοκρατία και κράτο δικαίου, αλλά καθίστε απόλυτα σαφέ ότι αυτό ε, για, η συμπεριφορά ειδική αποδεικνύει πως αγνοείται, παραγνωρίζεται πλήρως το κράτο δικαίου και δεν εφαρμόζεται πουθενά τις συνθήκε συνθήκες και τους κανόνε που έχουν, ε, που έχουν εισαχθεί. Θέλω να ακούσω την απάντησή σα. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας για το θέμα των αποσπάσεων των εργαζομένων. Είναι σαφές ότι η οδηγία για τις αποσπάσεις είναι μια πολύ περίπλοκη οδηγία και οι ιδέες τις οποίες εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του μετά από την εκλογή του η οποία θυμίζω έγινε με μια άνετη πλειοψηφία, είναι μια σωστή ιδέα αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Μπαρόσο. Θα πρέπει να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο η οδηγία αυτή ε, και να συζητηθεί ε, λεπτομερέστερα. Αλλά αυτό δεν έχει μπορέσει να γίνει μέχρι τώρα γιατί δεν ελέγχουμε απόλυτα ε, το περιεχόμενό της ακόμη. Δεν την έχουμε εφαρμόσει πλήρως. Από την άλλη να θυμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να υπάρξει κανένα εμπόδιο στη διακίνηση των εργαζομένων και, θα πρέπει, δεν θα, και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων να θυγούν. Το θέμα λοιπόν το οποίο πράγματι τίθεται πέρα από αυτά που λέει το κείμενο είναι η εφαρμογή τους και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος μπορεί να βρουν μια λύση στα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να χαίνουν. Είναι σαφές βέβαια ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται μια σε βάθος πολιτική συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο της οδηγίας. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω σε αυτή τη φάση τα χαρακτηριστικά τα οποία θα λάβει η συζήτηση αυτή. Υπάρχουν αρκετές αναλύσεις και αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Έχουν γίνει επαφές επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι φυσικά εξέφρασαν τις απόψεις τους και περιμένουμε ε, τις απαντήσεις ορισμένων άλλων εταίρων. Έχουμε αντιμετωπίσει με δυναμικό τρόπο το πρόβλημα και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε αυτόν τον πολιτικό δυναμισμό σχετικά τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την χρηματοδότηση 100% από κοινοτικά ταμεία. Γιατί υπάρχουν ορισμένες χώρες μέλη όπου είναι σαφής μια πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιου είδους μορφές χρηματοδοτήσεως. Θυμίζω ότι πλησιάζουμε στην χειμερινή περίοδο αυτό σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένες περιοχές και σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό ακριβώς κάναμε λοιπόν την πρόταση αυτή. Είναι μια πρόταση η οποία έχει σαν στόχο την απλούστευση της λειτουργίας του Ταμείου μέσω βέβαια της, του σεβασμού του κανονισμού του του κανονισμού λειτουργίας του. Βέβαια δεν έχει τύχει πλήρους υποστήριξης από το σύνολο των κρατών μελών και υπάρχει μια μειοψηφία στο Συμβούλιο η οποία μπλοκάρει τις προτάσεις μας. Σε αυτή τη φάση είναι αδύνατο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια νέα πρόταση, πρέπει να περιμένουμε. Και απλά προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Προεδρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να βρούμε μια λύση, μια λύση η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει αυτούς που αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Το τι μορφή θα πάρει αυτή η προσπάθεια δεν είναι σαφές. Υπάρχουν τρεις επιλογές ανοιχτές μπροστά μας. Στην φάση που βρισκόμαστε τώρα απλά συνεργαζόμαστε με την Προεδρία και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου να διαπιστώσω εδώ κάτι το οποίο ξέρετε. Ξέρετε ότι αυτός που δίνει λέμε κάτι γρήγορα στη χώρα μου δίνει δυο φορές περισσότερα από αυτόν που αργεί. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να έχουμε καθυστερήσει. Η κοινωνική κρίση είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτή και θα πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσες και όχι να αναζητούμε κάθε φορά την τελειότερη λύση η οποία θα αργήσει πολύ να βρεθεί. Πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με την Προεδρία, με την κάθε Προεδρία, να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, δηλαδή ένα συμβιβασμό. Σχετικά τώρα με την κοινωνική πολιτική και την αξιολόγηση ε, της αποτελεσματικότητας αυτής της ε, κοινωνικής πολιτικής, αυτό θα γίνει σε έφθετο χρόνο να διαπιστώσω όμως κάτι μαζί σας, ότι η Ευρώπη καταρχάς έχει διευρυνθεί, υπάρχουν πολλές νέες χώρες και το να συνεχίσει κανείς να έχει τα ίδια μέσα και τις ίδιες προσδοκίες για την πολιτική αυτή που είχε πριν από τη διεύρυνση είναι κάτι περίπλοκο. Ελπίζω όμως παρόλα αυτά ότι δεν μιλάμε για μια στασιμότητα. Μιλάμε για κάποια πρώτα βήματα πρόοδου, για την καταπολέμηση της φτώχειας Ξέρετε ότι έχουμε ήδη καταθέσει κείμενα που αναφέρονται στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε μιλήσει για τη φτώχεια και τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στην παιδική ηλικία. Αναφερόμαστε δηλαδή στις ανάγκες των παιδιών που ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες το έτος για την καλαπολέμηση της φτώχειας διακηρύχθηκε ακριβώς για να ενισχύσει τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε και να τις γνωστοποιήσει ακόμα περισσότερο και για την ισορροπία που θα πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μέσα και τα εθνικά μέσα, η ισορροπία αυτή είναι αγκυρωμένη στη συνθήκη θυμίζω. Η συνθήκη αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής με κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες καθορίζονται ακριβώς από την ίδια τη συνθήκη στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Προφανώς είναι πολιτικό το θέμα. Μπορεί κανείς να έχει ερωτηματικά για την ικανότητα με την οποία τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα και είναι ζητούμενο να δούμε αν πράγματι οι κανονισμοί ευρωπαϊκοί ορίζουν ένα σαφές πλαίσιο. Σχετικά τώρα για την ερώτηση που έφεσε η Λιθουανή συνάδελφος, ήδη έδωσα κάποιες απαντήσεις στα πλαίσια της απάντησης στην ερώτηση της κυρία Όταν μίλησα για αλλαγές στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Είπα ότι προσπαθούμε να αναζητήσουμε το ταχύτερο δυνατόν μια συμβιβαστική λύση. Λοιπόν, περνάω τώρα στο θέμα της εταιρείας Dell. Ακριβώς αυτό το Ταμείο Ρύθμισης για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Έκανε μια πρόταση η Ιρλανδική κυβέρνηση και το συζητήσαμε το θέμα, όπως συζητήσαμε και όλες τις προτάσεις οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν. Το Ταμείο αυτό προσαρμογής λοιπόν λειτουργήσε, εγώ επισκέφθηκα τη μονάδα παραγωγής, συζήτησα με τους υπευθύνους και τους εργαζομένους και διαπίστωσα ότι οι εργαζόμενοι πράγματι θεώρησαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήταν κάτι το πολύ σημαντικό για αυτούς, ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια. Για το Ταμείο Προσαρμογής Ξέρετε ότι ε, τώρα έχει αρχίσει να λειτουργεί αυτό το ταμείο. Ξέρετε ότι το συγκεκριμένο αυτό ταμείο θα αποκτήσει μια διάσταση στο μέλλον πολύ πιο σημαντική. Για το 2009 υπήρξε μάλιστα και μια αλλαγή στους κανονισμούς η οποία αποφασίστηκε από κοινού, θυμίζω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή ήταν μια κομβική στιγμή στην εμπειρία που είχαμε. Τώρα, το 26.000 που βοηθήθησαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Προσαρμογής της Συνέπειες Παγκοσμιοποίησης. Κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλος αριθμός. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε φορά που συζητώ με τους δικαιούχους, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς τους ανθρώπους και ο αριθμός αυτός φυσικά οφείλει να μεγαλώσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Αυτή τη φορά θα είμαστε πιο αυστηροί με το χρόνο για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο ο κύριος Μπιαρή και μετά η κυρία Καρίμα Ντέλη. Κύριε Επιτροπέ, έχω τρεις ερωτήσεις. Θα δώσετε στο Ευρωπαϊκό Εργασιακό Συμβούλιο την δυνατότητα να μπλοκάρει τις προτάσεις απόλυσης, μια και οι προτάσεις αυτές έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων ή την καλύτερη αμοιβή των μετόχων. Η εταιρεία Dell ε, ήδη αντιμετώπιζε δυσκολίες, αλλά το πρόβλημα ήταν περισσότερο η μετεγκατάστασή της. Ήταν σχέδιο μετεγκατάστασης αυτό. Ε, εκφράζετε την ικανοποίησή σας για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία. Βέβαια, δημιουργείται ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων. Θα εξετάσετε τη δυνατότητα μιας εναρμόνισης προς τα πάνω των ε, μισθολογικών επιπέδων και των επιπέδων κοινωνικής προστασίας. Είστε έτοιμος να διευκρινίσετε τον όρο υπηρεσίες κοινοφελής ή γενικού συμφέροντος. Η κυρία Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένη με την παρατήρησή σας λίγο πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει γίνει μια μελέτη που ε, διαπιστώνει ότι 118 εκατομμύρια είναι οι φτωχοί στην Ευρώπη. 118 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν φτώχεια και επισφαλή απασχόληση. Και ε, ιδιαίτερα τι κατάσταση πλήττους νέους, τις γυναίκες, έχουν προβλήματα στέγασης, πρόσβαση στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας κτλ. Προβλέπετε φέτος κάποιες δράσεις για τις ευπαθέστερες αυτές ομάδες του πληθυσμού και ποιοι είναι οι στόχοι σας. Μιλήστε για κάποια κείμενα για την προστασία των παιδιών, αλλά ποιοι είναι οι στόχοι σας προκειμένου να μειώσετε τις ανισότητες. Ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία. Γιατί για να μειώσουμε τις ανισότητες θα πρέπει να μειώσουμε τα χάσματα μεταξύ των εισοδημάτων. Γιατί ακόμη και σήμερα έχουμε διευθυντικά στελέχη που λαμβάνουν παχυλές αποζημιώσεις ενώ προηγουμένως έχουν απολύσει και έχουν βγάλει στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους. Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να προτείνει υποχρεωτικούς κανόνες προκειμένου να περιορίσει τα εισοδήματα και να ε, προβεί σε μια καλύτερη ανακατανομή του πλούτου. Σας ευχαριστώ κυρία Πασκάλ Γκρούνη και μετά ο κύριος Αλεχάνδρο Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την οδηγία για το ωράριο εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νέα πρωτοβουλία, γιατί δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία της νέας οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τι ανισότητε σε θέματα κοινωνική προστασία, πώ ε, σκοπεύετε να τι ε, γεφυρώσετε, γιατί έτσι είναι που δημιουργείται στρέβλο ανταγωνισμού και επιτείνονται οι ανισότητε μεταξύ των Ευρωπαίων. Τι γίνεται με την ισότητα των δύο φύλων, ποιε είναι οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και τι γίνεται με την κοινωτική στρατηγική σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασία. Ο κύριο Σέρκα. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, Επίτροπο. Έχω ένα σύντομο σχόλιο και τρεις ερωτήσεις. Μιλήσατε για την κρίση της Ευρώπης χαρακτηρίζοντας την ως κρίση αξιών. Δυστυχώς όμως μείναμε ορφανοί από την ανάλυση σας. Γιατί ακούσαμε για την οικονομική κρίση, ακούσαμε για τη δημογραφική κρίση. Για τις αξίες όμως που είπατε ότι χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή κρίση δεν ακούσαμε κουβέντα. Θα πρέπει να βρούμε τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών το χάσμα που υπάρχει, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το ευρωπαϊκό σχέδιο και όραμα. Δυστυχώς ούτε και εσείς, ούτε και ο Επίτροπος, ε, ούτε και εσείς, ο Πρόεδρος Μπαρόζο μας πείσατε. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, καταρχήν, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Ο πρόεδρο Μπαρόζο, όμω, είπε στη σοσιαλιστική ομάδα ότι δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα εφαρμογή, αλλά και πρόβλημα ερμηνεία εγώ θα έλεγα ότι μάλλον ένα πρόβλημα σχέσεων, σύνταξη της οδηγίας υπάρχει. Αυτή είναι η γνώμη όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας. Πιστεύετε ότι είναι πρόβλημα ερμηνείας ή είναι διοικητικό πρόβλημα εφαρμογής αυτό που υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για το ωράριο εργασίας. Φαίνεται ότι η θέση σα πάει από τη θέση όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Πρόεδρου Μπαρόζο. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να θέσει τέρμα στην αποδυνάμωση τη ασφάλεια των εργαζομένων. Και ο Πρόεδρο Μπαρόζο μα υποσχέθηκε μία μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων. Εσεί μα είπατε ότι θα γίνει μελέτη επιπτώσεων, αλλά όχι κοινωνικών επιπτώσεων. Δυστυχώ οι κοινωνικέ συνέπειε φαίνεται ότι ε, εξαφανίστηκαν από την πρόταση για τη μελέτη του αντικτύπου. Επίσης, Μα υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ισχυρό μηχανισμό για τι κοινοφελεί υπηρεσίε ή τι ε, υπηρεσίε ε, γενικού συμφέροντο. Παραλείψατε τελείω από την ομιλία σα αυτή την πρόταση. Μήπω διαφωνείτε με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα έκανε τη σχετική υπόσχεση. Ευχαριστώ. První eh, eh, byla Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια ερώτηση που αφορούσε την εναρμόνιση προς τα άνω. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω και να επαναλάβω ότι η Επιτροπή και οι Επίτροπη είναι υποχρεωμένοι να ε, ακολουθούν τις επιταγές της ενισχύ συνθήκης. Και Ευρώπη σημαίνει πρόοδος. Η Επιτροπή ακολουθεί εκ του σύνεγγης τις κοινωνικές προόδους, την εξέλιξη στα κοινωνικά θέματα. Και σε κάθε μία από τις αποφάσεις μας, πάντοτε γνώμονα έχουμε την ικανοποίηση των της ανάγκης της συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων αγορών εργασίας, δηλαδή να μην υπάρξει ζήτημα ε, του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας μεταξύ των μελών. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερη μέρημνα και ε, προσπάθειες εκ μέρους μας. Τα όσα αναφέρατε για τη φτώχεια και για τις ε, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τα έχουμε εμείς προβάλει, η Επιτροπή. Βλέπουμε ότι δεν έχει όντως αυξηθεί η φτώχεια, αλλά δεν έχει ούτε μειωθεί. Και έτσι πρέπει να δούμε σε μια κρίση τόσο βαθιά τι ενδεχόμενα υπάρχουν να αυξηθεί η φτώχεια. Και βέβαια θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να λάβουμε τα καταλληλότερα μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε θεσπίσει εξάλλου το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας, προσπαθώντας να βρούμε τα καταλληλότερα μέτρα για μια καλή ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουμε διατυπώσει ε, τις θέσεις Επιτροπής σε έγγραφο με τίτλο «Ενεργός ενσωμάτωση», «Ενεργή ενσωμάτωση», ε, όπου μιλούμε για ελάχιστο εισόδημα, για αποφύγη των διακρίσεων και για στεναρές κοινωνικές παροχές που θα προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας. Για τη μείωση του χρόνου εργασίας που ανέφερε ο κ. Σέρκας, θα ήθελα να πω ότι η πρώτη θέσή μας, προσπάθεια μας, είναι να επιτύχουμε πρόοδο στο σημείο αυτό. Το σχέδιο θα είναι ένα σχέδιο, ένα εγχείρημα περίπλοκο, δεν θα είναι εύκολο δηλαδή να τοποθετηθεί κανείς. Ε, θα πρέπει να βρούμε μία λύση συμβιβαστική σωστή που να σταθμίζει και την ανάγκη κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων σωστά. Κάτι που ξέρουμε, όπως άλλωστε το έπαιξε τα τελευταία πέντε χρόνια, ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο τα άλλα ερωτήματα που μου απευθύνθηκαν. Έχουν διατυπωθεί με πολύ ε, εύγλωτο τρόπο. Ερωτήματα που θυμίζουν, θα έλεγα, δίκη. Θα ήταν αντίστοιχα με αυτά που θα μου απίθενε ο εισαγγελέα, αν θέλετε, στην περίπτωση κάποιας διαφοράς ε, δικαστικής ή αγώνα δικαστικού. Εγώ φυσικά θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στην ερμηνεία και όχι στη διαφορά, γιατί και η ερμηνεία ασφαλώς επηρεάζει τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων. Και εδώ έχουμε ένα πολύ περίπλοκο ε, σχηματισμό, ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον. Ζητήματα τα οποία όμως θα πρέπει να συζητηθούν είναι επί η ε, μελέτη των επιπτώσεων που ιδιαίτερα θα πρέπει να εξετάσει βέβαια τις κοινωνικές επιπτώσεις και το ότι αναφέρθηκαν ενδεχομένω σε ένα πιο γενικό ή ανώτερο αν θέλετε επίπεδο δεν σημαίνει ότι δεν θα ε, αναπτύξουμε μελέτη επιπτώσεων κοινωνικών του Το ότι δεν αναφέρθηκα ρητά στις, στη μελέτη των οικολογικών επιπτώσεων δεν σημαίνει ότι δεν θα σεβαστούμε τα ζητήματα, θα γίνει μελέτη των οικολογικών επιπτώσεων. Τώρα για την οδηγία περί ε, υπηρεσιών κοινή ωφελία, όπου θεωρώ ότι η αλλαγή της νομοθεσίας θα μπορούσε να προσφέρει θετικά αποτελέσματα, ωστόσο Οφείλω να ομολογήσω ότι η θέση την οποία εγώ πρεσβεύω δεν έχει γίνει δεκτή ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι, δεδομένου ότι ε, θεωρούνται ύπατη σημασία σημασία αυτές οι υπηρεσίες, προσπαθούμε, ξεκολουθούμε τις προσπάθειες για να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ παρέμβασης ή διαβήματος σε νομοθετικό επίπεδο, νομοθετικού τύπου ή κάποιες άλλες λύσεις. Θα ήθελα ίσως να δώσω και άλλες απαντήσεις, αλλά βλέπω ότι η κυρία Πρόεδρος με κοιτάει με πολύ αυστηρό ύφος και θα πρέπει να περιμένω μια ερώτηση για να δώσω την απάντηση. Ευχαριστώ Κύριο κύριος Ντεράικλερ και ο κύριος Κλάρκ. Ε, ο και κοιτάω αυστηρά, απλώς ο κανόνας πρέπει να τηρείται. Αυτά, απλά πράγματα. Ο κύριο Ντεράικλερ. Ευχαριστώ. Είπατε κύριε Επίτροπε θέλετε να βοηθήσετε τους ανέργους. Και κατόπιν μιλήσατε για ρύθμιση, για οδηγίες, για πρωτοβουλίες, για διαθροδοτικές αλλαγές και τα υπόλοιπα της κοινωτικής ορολογίας. Εγώ λαμβάνω όλο και περισσότερα γράμματα από εκλογής μου που απαντούν στο ερώτημα ποιος ε, είναι ο αντίκτυπος της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι απαντήσεις τους ξεκινούν από ότι είναι βάσανο και ε, δημιουργούν χρονοτριβές έως ε, οδηγούν σε επιδείνωση της κατάστασης των επιχειρήσεών τους, σε απολύσεις, σε απώλειες κτλ. Βλέπετε ότι είναι ευρύ το φάσμα των απαντήσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει απασχολούν σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μια τέτοια δυσμενή γνώμη για την κοινωτική νομοθεσία είναι πολύ κακά μαντάτα. Στη συνδιαλλαγή για το οδηγία του χρόνου εργασίας που κατέληξε σε αποτυχία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η αποτυχία σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκε από το γεγονός ότι πριν από πέντε χρόνια, όταν μόνο λίγες χώρες ήθελαν ε, αυτοεξαίρεση από την ε, οδηγία για το χρόνο εργασίας, ε, οι χώρες από πέντε που ήταν στην αρχή που ήθελαν αυτοεξαίρεση έγιναν 15 από τις 27. Αυτό θα πρέπει να σας δίνει ένα μήνυμα ότι ο κόσμος αυτό που θέλει να συνεχίσει τη ζωή του και να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς καμία επιρροή και επίδραση από την κοινωτική νομοθεσία. Ο κύριος Χάντελ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δύο σύνολα, αν θέλετε, ερωτήσεων. Το πρώτο σχετικά σύντομο. Μια απλή ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι η αυτονομία ως προς τον προσδιορισμό, η ανεξαρτησία ως προς τον προσδιορισμό των συλλογικών συμβάσεων ε, θα έχει θέση στο ευρωπαϊκό ε, κοινωνικό γίγνεσθε και αν όχι γιατί. Και δεύτερον, στα θέματα που έθιξε και ο κύριος Τόμας ε, Μαν ε, για το ζήτημα της Όπελ, θεωρώ ότι η ερώτηση ήταν ε, και η απάντηση ήταν μάλλον ρητορικού χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να σας αφήσω να ξεφύγει τόσο εύκολα και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για μια άλλη υπόθεση που είχε ιδιαίτερη απήχηση. Η Ντέλ αποφάσισε να κλείσει μια επιχείρηση στην Ιρλανδία ανησυχούν πολλοί συνάδελφοι. Βοηθάμε 14,8 εκατομμύρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση έτσι ώστε να βοηθήσουν του συναδέλφου, του εργαζομένου να βρουν εκεί κάποιε άλλε λύσει. Το, ότι πηγαίνει όμω η Ντέλ όχι στην Κίνα αλλά στην Πολωνία ασφαλώς αποτελεί κέρδο για τους ανέργου τη Πολωνία που θα βρουν κάποια θέση εργασία. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς προσφέρει πάλι την υποστήριξή της με 48,5 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Εάν μέσα σε τρία χρόνια η Ντέλα αποφασίσει να ξανακλείσει το εργοστάσιο, αυτή τη φορά στην Πολωνία, θα δραστηριοποιηθεί και πάλι το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση για να δώσουμε πάλι ικανοποίηση στι δύσκολε καταστάσει που θα προκύψουν εκεί. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν πάει η Ντέλ στη Νότια Ιταλία, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει βεβαίω και του ανέργου τη Νότια Ιταλία, ευκταίων. Πάλι θα τους δώσει 50 εκατομμύριο παραδάκι. Μήπως λοιπόν στην Όπελ εφαρμόστε διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Δεν θα έπρεπε κάποιος ο οποίος κάνει τέτοιες κινήσεις το τι εγκαταστάσεις του να έχει αντί για έπαινο κάποιο είδους κύρωση. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά μια και μας περιορίζει ο χρόνος θα περιοριστώ σε μία μόνο. Καταρχήν θα επανέλθω στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Είδατε πόσε ερωτήσει υπευλήσα και καταλάβατε τι σύγχυση υπάρχει και παρεξηγήσεις. Όταν ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε στους σοσιαλιστές, είπε ξεκάθαρα ότι θα υπέβαλε έναν εφαρμοστικό κανονισμό, αφήνοντας ανέγκυχτη την οδηγία. Αλλά άλλο οδηγία, άλλο κανονισμός η οδηγία, γιατί η οδηγία είναι για την απόσπαση των εργαζομένων, αφήνει περιθώριο ελιγμών και ερμηνεία στα κράτη-μέλη. Γιατί λέει ότι τα κράτη-μέλη δίνανται. Ενώ ο κανονισμό ε, είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη και προβλέπει με σαφήνεια τι οφείλουν να κάνουν. Πώ θα συνδυαστούν λοιπόν μια οδηγία με ένα κανονισμό. Κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια θα είναι η φύση αυτού του, ε, του νομοθετήματος πριν ε, μιλήσει ο Μπαρόζο ή κάπως πρόλαβε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι δηλώσει του. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο, θα ήθελα να επανέλθω στην υπόθεση τη ΔΕΛ. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι από άποψη Ταμείου Παγκοσμιοποίηση ε, υπάρχει μια λογική που ακολουθείτε. Αλλά ω ε, μέλο ενό συλλογικού οργάνου δεν μπορείτε να αγνοείτε, δεν μπορεί η δεξιά να αγνοεί πει η αριστερά. Και όταν εξετάζουμε το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την εταιρεία Dell, ε, καταλήγω σε τέσσερα διδάγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνόησε και στήριξε μία διαδικασία μετεγκατάστασης χάρη στην κινητοποίηση του Ταμείου παγκοσμιοποίηση αφενό και χάρη στην άδεια κρατικών ενισχύσεων αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στην επιχείρηση Dell να εξαγγείλει ταυτόχρονα την εξαγορά του συστήματος Perot, κάτι που επέτρεψε στην ε, επιχείρηση Dell να κερδίσει πολλά δολάρια και να ενισχύσει τη μετοχή της. Τρίτο δίδαγμα στην επιχείρηση αυτή κανένα από τις, καμία από τις αρχικές αρχές του σχεδίου ανάκαμψης δεν τηρήθηκε και κυρίως ο σκοπός διαφύλαξης των θέσεων απασχόλησης και διαπιστώσαμε ότι απαιτήθηκε η επιστροφή της εγγύησης ε, για τις εγκαταστάσεις στην Τέλη στην Ιρλανδία. Γνωρίζουμε τη λογική του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και στηρίζουμε αυτή τη λογική. Είναι απαράδεκτο όμως η εφαρμογή αυτής της λογικής να οδηγεί σε μια τέτοια κατάσταση όπου σε τελική ανάλυση τα κονδύλια του φορολογούμενου, τα χρήματα του φορολογούμενου ευνοούν μια μετεγκατάσταση και γεμίζουν τις τσέπες του Αμερικανού μετόχου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόγνω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία πως έχουν τεράστια σημασία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δε πλειονότητα των ευρωπαϊκών διατάξεων διευκολύνει ως προς τον διοικητικό γραφειοκρατικό φόρτο μια επιχείρηση η οποία παραδείγματι δρά στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να υποφεληθεί της αρχής της αναγνώρισης, αντί, της αναγνώριση. αναγνώρισης, δηλαδή για 27 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια μπορεί να δρά βάσει ενός νομοθετικού πλαισίου μια μικρομεσαία επιχείρηση. Η Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση για ένα νομοθέτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ε, τα όρια πληρωμών που ε, είναι πιο ευνοϊκά για τις μικρομεσαίες σε σχέση με τις ε, μεγαλύτερων διαστάσεων επιχειρήσει. Γενικά, δηλαδή, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κάθε μας πρωτοβουλία, το better regulation και ό,τι άλλο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίζουμε το γραφειοκρατικό άχθο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά, ο καθένας μπορεί να προβάλλει κάποια λεπτομέρεια από εδώ ή από εκεί και να συζητήσουμε κάποια λεπτομέρεια, αλλά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ρητά να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, αναγνωρίζεται η σημασία, η αξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εν προκειμένου υπογραμμίζω ότι είχα πολλές επαφές με εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των κοινωνικών ε, εταίρων και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι και οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η, ε, η ικανότητα για ανάπτυξη υπερεθνικού διαλόγου. Έγινε λόγος για την ΟΠΕΛ, έγινε λόγος για την Dell. Διαπιστώνεται όλο και οι περισσότερες συναλλαγές αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μέσα στα όρια ενός κράτους μέλους. Εν προκειμένου λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και αυτός είναι ο κύριος μας προσανατολισμός για την Όπελ. Είχα την ευκαιρία ε, μετά το, την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτο ε, στην Τσεχική Δημοκρατία και με τα καθήκοντα που είχα εκεί ω υπουργό να αναπτύξω δραστηριότητε αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή να συμμετάσχω και εγώ στι δραστηριότητε αναδιάρθρωσης. Και ήθελα να πω εδώ ότι στην ε, σημερινή μα κατάσταση δεν είναι σε θέση βέβαια να επεκταθώ σε όλε τι λεπτομέρειε. Υπάρχουν κάποιε βασικέ αρχέ. Η βασική αρχή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για τον αυστηρό σεβασμό κάθε κανόνα και την ε, αποτελεσματική ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου. Η Dell αποφάσισε τη μετακίνηση της επιχείρησης το 2005 ή 2006. Ασφαλώς λοιπόν θα πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Το ότι δίνει την έγκρισή της για την ενίσχυση προς την πολωνική κυβέρνηση η Επιτροπή είναι σαφές. Στηριζόμαστε σε κανόνες ενισχύει και τηρούμε απόλυτα τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μόνη προσέγγιση που μπορούσαμε να έχουμε στην τελευταία ανάλυση. Για δε το Ταμείο Προσαρμογής δεν ε, οφείλεται στη λειτουργία του Ταμείου Προσαρμογής ε, η απόφαση σχετική με την ΤΕΛ, γιατί έχει ληφθεί δύο χρόνια πριν από τη θέση λειτουργία του Ταμείου Εισαγωγής. Πάντως θα ήθελα να υιοθετήσω θα ήθελα να επισημαίνω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ε, μονοσήμαντη, μια λιγότερο μονοσήμαντη προσέγγιση. Είναι πολλά τα στοιχεία που ε, μας οδηγούν στη λήψη μίας απόφασης σε σχέση με την μετακίνηση μιας εταιρείας, μιας επιχείρησης από τη μια περιοχή στην άλλη. Είναι πολλά τα δεδομένα, περίπλοκη εικόνα που σχηματίζεται, ο οικονομικός κύκλος, η οικονομική ζωή είναι τόσο περίπλοκα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα μερικές φορές και πρέπει όλα αυτά βέβαια να κρίνονται με βάση την οικονομική λογική και βέβαια ε, ορθώς νοούμενες κοινωνικές πρόοδους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην οδηγία από τη μία και στους κανονισμούς από την άλλη και νομίζω ότι η συζήτηση επί της ουσίας είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον. Στην προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε αρκετά σημεία τα οποία ελπίζω ότι στο μέλλον θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ελπίζω να έδωσα τις απαντήσεις που θα θέλατε. Κρίστιανσεν και μετά η κυρία Μωρά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που μας επισκέπτεται. Είναι αλήθεια ότι στα πλαίσια της κρίσης στην οποία ζει η Ευρώπη πολλοί φοβούνται για τη μονιμότητα των θέσεων απασχόλησης τις οποίες κατέχουν. Ο ανταγωνισμός γίνεται όλο ένα και πιο σκληρός. Ο ανταγωνισμός αυτός όμως θα πρέπει να σέβεται ορισμένα, θα έλεγα, ορισμένα στιγμία. Δεν μπορεί να δεχόμαστε στην εισαγωγή απλά εργαζομένων από το εξωτερικό μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότεροι. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν ιδιαίτερα σε επίπεδο αμοιβών, μισθών και αμοιβών. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι πάντα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει κάποια επιπλέον μέτρα όταν τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τους κανόνες. Η κυρία Μωρά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε προηγουμένως στις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφιλίωση της προσωπικής ζωής με την επαγγελματική ζωή, της οικογενειακής μάλλον με την επαγγελματική δραστηριότητα. Τι μέτρα μπορείτε να πάρετε για να αντιμετωπίσετε την ανισότητα στις σταδιοδρομίες ανδρών γυναικών, τις ανισότητες σε επίπεδα συνταξιοδότησης, για να μην αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών και επίσης στο τι μέτρα θα ληφθούν για τις γυναίκες μόνες οι οποίες θέλουν να ασκήσουν τις, την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Είπατε ότι η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αναφερθήκατε και στις εξελίξεις προς μια οικονομία φτωχή σε διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό περνάει μέσα και από την προσαρμοστικότητα πράγματι των εργαζημένων. Πώς μπορούμε εμείς να συνδυάσουμε την κινητικότητα την επαγγελματική με την γεωγραφική κινητικότητα ενώ ταυτόχρονα τα θέματα της κατάρτισης και τα θέματα της πιστοποίησης των γνώσεων των εργαζομένων είναι διαδικασίες στατικές και θα πρέπει να τις καταστήσουμε με κάποιο τρόπο πιο γρήγορες και αποτελεσματικές. Η κυρία Ράπτη παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας. Ε, είπατε προηγουμένως ότι αισθάνεστε πως οι ερωτήσεις που γίνονται σε αυτή την, εδώ την αίθουσα προς εσάς θυμίζουν δίκη. Επειδή αναφέρατε διάφορες σοφές κουβέντες που λέγονται στην πατρίδα σας, επιτρέψτε μου να σας πω και εγώ μία-δύο κουβέντες που λέγονται στη δική μου πατρίδα, την Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν λέμε ότι όταν κάποιος αισθάνεται πως του επιτίθενται όλοι, είναι ίσως καιρός να δει τι έχει κάνει λάθος ο ίδιος. Θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Μιλήσατε για ήτες και νίκες. Θέλετε να μου πείτε τι θεωρείτε ήτες και τι νίκες και αν θεωρείτε ότι οι ήτες αυτές και οι νίκες αυτές ταυτίζονται με τις νίκες και τις ήτες που θεωρούν οι εργαζόμενοι. Και κάτι τελευταίο. Το τελευταίο είναι εάν κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσετε μία αξιολόγηση της αναθεωρημένης κοινωνικής ατζέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εσαϊά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπε. Όπως είπατε κύριε Επίτροπε, αυτό που έχει σημασία είναι το τι μέτρα θα πάρουμε για τη στήριξη της απασχόλησης και σε αυτό θα πρέπει να εμείνουμε όλοι. Να πω εδώ ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται. Και ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες μας οι οποίοι έχουν επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες μοιράζονται θα έλεγα σε διαφορετικές χώρες. Έχουν ένα παρελθόν επαγγελματικό σε διαφορετικές χώρες. Και τι γίνεται ακριβώς με τις συντάξεις τους όταν έχουν εργαστεί σε δύο, τρεις ή τέσσερις χώρες. Πού γίνονται σεβαστά τα βασικά τους δικαιώματα, τα συνταξιοδοτικά. Τι κάνετε εσείς σαν Επιτροπή για να διευκολύνετε την συνταξιοδότηση των πολιτών αυτών που είναι χαμένοι στο μέανδρο των γραφειοκρατικών διαδικασιών πολλών κρατών μελών μερικές φορές. Βοηθήστε λοιπόν τους εργαζομένους. Βρείτε μέτρα. Ο κύριος Τσάμπα Όρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι δύσκολα τα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα. Δεν ξέρω αν πράγματι μιλάμε για το παρελθόν ή για το μέλλον. Αν μιλάμε για το παρελθόν θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά τον κύριο Σπίτλα Πρέπει να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν ένας από αυτούς ε, τους οποίους όταν του ζητήσαμε να μας συναντήσουν ήλθε εδώ, συζήτησε μαζί μας ο κύριος Σπίτλα και επέδειξε θετικό πνεύμα, πνεύμα συνεργασίας και θα θέλαμε να συνεχιστεί. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι ξεκάθαρα υπέρ της επαναδιατύπωσης της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Αντίθετα, μέχρι τώρα δεν ακούσαμε και πάρα πολλά για τις λεγόμενες νέες θέσεις απασχόλησης και για τις λεγόμενες ατυπικές μορφές απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά σε βάθος. Λοιπόν, νέες μορφές απασχόλησης, ατυπικές μορφές απασχόλησης, ανάπηροι στην απασχόληση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους ανάπηρους εργαζομένους. Κάντε κάποια σχόλια και για την περίπτωση αυτή κύριε Σπίτλα. Ανάπηροι εργαζόμενοι. Pokud je otázky eh, rovnosti nebo respektive eh, odměňování nebo σχετικά με τα θέματα της ισότητας αμοιβή για ίση εργασία είναι σαφές ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ορισμένα πράγματα από κοινού πρώτα. Υπάρχουν πολλές φορές διαφορετικές αμοιβέ για την ίδια περίπου εργασία στο εσωτερικό των ιδίων των χωρών. Επίσης υπάρχουν και σημαντικές διαφορές στον έλεγχο της παραγωγικότητας της εργασίας. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί δείκτες, πολλοί παράγοντες οικονομικοί και κοινωνικοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στις νέες χώρες υπάρχουν χαμηλότερες αμοιβέ, αλλά είναι φυσικά και χαμηλότερη η παραγωγικότητα. Η σχέση λοιπόν ε, αμοιβή και παραγωγικότητα είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω, έχει περιορισμένες δυνατότητες για να επηρεάσει το συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά τις δυνατότητες τις οποίες έχει τις εκμεταλλεύεται πιστεύω πλήρως και στα πλαίσια της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και στα πλαίσια του κοινωνικού ευρωπαϊκού διαλόγου. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τον εναρμονισμό είναι ακριβώς ε, αυτός ο κοινωνικός ευρωπαϊκός διάλογος και νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των μέσων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όσα και αν είναι αυτά και όσο λίγα και αν είναι. Και αυτό ισχύει και για την οδηγία, για την απόσπαση των εργαζομένων και κυρίως να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με την ισότητα εργασίας και αμοιβής. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια ανακοίνωση ε, με συγκεκριμένο στόχο την ισότητα ευκαιριών. Προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Είχαμε ορισμένα επιμέρους στοιχεία επιτυχίας και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει επίσης να πω ότι στα πλαίσια αυτής της συζήτησης που γίνεται εδώ από τη μία εγώ και από την άλλη εσείς κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, νιώθω άνετα, νιώθω ιδιαίτερα άνετα. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι επίπεδου, με βοηθά να καταλάβω ορισμένα πράγματα, με διαφορετικό τρόπο ίσως, δεν συμφωνώ φυσικά σε όλα όσα ακούω, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι είμαι ανάμεσά σας σήμερα και συζητάμε. Οι αντιδράσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε, ε, Απλά χρησιμοποίησα ίσως ε, κάποια λόγια που είπε και ο κύριος Σέρκας με λίγο διαφορετικό τρόπο. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια, ότι η συζήτηση η οποία προηγήθηκε ήταν ζωηρή και νομίζω χρήσιμη και για τους μεν και τους δε. Με ρωτήσατε επίσης το τι εγώ θεωρώ σαν επιτυχές αυτά τα οποία έχω κάνει. Αυτά θα το κρίνουν οι πολίτες. Ε, η οδηγία σαν παράδειγμα για την... Για την ενδιάμεση προσωρινή απασχόληση. Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει έχουν θεωρηθεί επιτυχή από όλε τι πλευρέ και θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Η ενίσχυση των συμβουλίων, των εργασιακών συμβουλίων. Ε, νομίζω ότι και εκεί έχει υπάρξει ε, ένα βήμα προόδου. Προφανώς τίθεται ε, το θέμα να κρίνει κανείς αν αυτά τα βήματα προόδου είναι επαρκή. Πολλοί μπορεί να έχουν αμφιβολίες γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει. Και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου έχουμε οδηγηθεί, σας θυμίζω, και ε, σε οδηγίες πιο επιμέρους όπως οι εργασίες στον χώρο της ναυτιλίας, η εργασία μάλλον ε, των ε, ναυτικών. Νομίζω ότι και αυτά είναι θετικά βήματα. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, να ισχυριστεί ότι θα έπρεπε να πάμε πιο μακριά ακόμα, να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Συμφωνώ μαζί σας. Πάντως έχουμε κάνει βήματα θετικά, βήματα επιτυχίας. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και γι' αυτό ακριβώς είμαι εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για τις λεγόμενες ατυπικές μορφές απασχόλησης ή νέες μορφές απασχόλησης. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και συμπεριλαμβάνονται και στην Πράσινη Βίβλο. Ο κύριος Τσάμπα Όρη μας μίλησε και για ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία γιατί θα έλεγα ο χαρακτήρας της αγοράς εργασίας είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να αλλάξει μέσω της προσπάθειας βελτίωσης των, της προστασίας των εργαζομένων και βελτίωσης και της λειτουργίας των κοινωνικών ε, συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ε, προφανώς θα συζητηθούν στο μέλλον. Ειδικά για τους αναπήρους. Το θέμα τις σχέσεις αναπήρων και εργασίας και των συνθήκων εργασίας των αναπήρων νομίζω έχει σχέση και με την οδηγία για την έλλειψη διακρίσεων. Νομίζω ότι έχουμε διατυπώσει ορισμένα κείμενα τα οποία είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένα που μπορούν να βοηθήσουν τους άμεσα ενδιαφερομένους και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να υπάρξουν ε, προσπάθειες εναρμόνισης σε συγκεκριμένους τομείς όπως οι κανόνες για τα συνοδά πρόσωπα σαν παράδειγμα όταν αυτό χρειάζεται ε, ή για τις συνθήκες για την μετακίνηση των αναπήρων στις ιδεοδρομικές μεταφορές ε, και της σήμανσης η οποία απαιτείται. Εκεί πρέπει να υπάρξουν μέτρα ενιοποίησης θα έλεγα και εναρμόνισης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ε, διαφορετικά συστήματα στις διάφορες χώρες. Εδώ έχουμε από τη μία τον κανονισμό 883 σχετικά με την μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Μετά από προσπάθειες οι οποίες κράτησαν 10 χρόνια απλοποιήσαμε τον κανονισμό και προσαρμοστήκαμε θα έλεγα στις λεγόμενες σημερινές ανάγκες. Πρόκειται όμως για μια προσπάθεια η οποία δεν έχει τερματιστεί, πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία τολμώ να πω δεν θα τερματιστεί ποτέ, συνεχώς θα αναζητούνται βελτιώσεις. Μια δεύτερη προσπάθεια την οποία κάναμε και εκεί αποτύχαμε. Αποτύχαμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό ήταν αρνητικό για τους ίδιους τους εργαζομένους είναι ότι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε με την οδηγία της μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε επίπεδο επικουρικών συντάξεων. Είναι περίπλοκο να σας το εξηγήσω, αλλά παρόλα αυτά ε, τα θέματα είναι σχετικά περίπλοκα σε επίπεδο πρωτογενών συστημάτων συνταξιοδοτικών, σε επίπεδο επικουρικών συνταξιοδοτικών συστημάτων τα συστήματα είναι εκτός ελέγχου σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που παρατείνατε το χρόνο σας ε, στη συνεδρίαση για να προλάβετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι τα καταφέρατε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε την αίσθηση ότι ήσταν στο εδόλιο προς σε ένα δικαστήριο. Ήταν μια συνηθισμένη ανταλλαγή απόψεων και ερωταπαντήσεων μεταξύ Ευρωβουλευτών και Επιτρόπου. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας. faire d'elle. Oui, oui. Oui, parce que ce n'est Bien, chers collègues, vous comprenez les raisons qui nous ont. Ξεφύγαμε λίγο από το ωράριο της ημερήσιας διάταξής μας. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, δεν συνηθίζω να παραβαίνω το χρονοδιάγραμμά μας ειδικά για τα ωράρια των ψηφοφοριών, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του Επιτρόπου για να προλάβουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. Και τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Προχωρούμε στο σημείο 7 της σας διάταξης που προβλέπει ψηφοφορία της έκθεσης Bauer για το ωράριο εργασίας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών είχαμε κάποιες δυσκολίες. Ε, όσοι έχουν ξεχάσει την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας τους θα πρέπει να το δηλώσουν. Δεύτερον, όσοι έχουν ε, κάποιες ε, παλιές κάρτες ψηφοφορίας, μάλλον δεν θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν. Τρίτη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε ότι κάθε κοινοβουλευτική ομάδα δεν ξεπερνά τον αριθμό των ψήφων που δικαιούται και δεν ε, έχει φέρει περισσότερους βουλευτές για να ψηφίσουν. Καταρχήν, ποιοι δεν έχουν τις νέες κάρτες ψηφοφορίας. Και μάλιστα δίνω εγώ το κακό παράδειγμα. Ποιοι έχουν ξεχάσει τις νέες κάρτες. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν μαζί τους τις κάρτες ψηφοφορίας. Οπότε κάθε φορά αυτοί οι τρεις συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνουν για το πώς ψηφίζουν. Ας κάνουμε μια δοκιμή καταρχήν. Για να εξακριβώσουμε ότι λειτουργούν όλες οι κάρτες. Και φυσικά να αποφύγουμε υπερβολική εκπροσώπηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Alors, euh, le vote test. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ παρακαλώ θα πρέπει να αφαιρέσει δύο ψήφους. Θα πρέπει να διώξει δύο μέλη του. Κύριε Ορή, αποφασίστε εσείς ποια θα είναι τα θύματα. Θα τα βρούμε μεταξύ τους. Έχουμε και άλλη δυσκολία όμως, τέταρτη. Δεν ξέρω ποιος, αλλά κάποιος μπλόκαρε το σύστημα εδώ. Ο κύριος Σέρκας. Κυρία Πρόεδρε, το ηλεκτρονικό σύστημα κανονικά πρέπει να μας διευκολύνει την ζωή, γιατί φαίνεται ότι μας την ε, περιπλέκει. Και αν έχουμε μόνο μια ψηφοφορία, γιατί να μην ψηφίσουμε διανατάσσεω της χειρός και χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, αυτά είναι τα προβλήματα, τα αρνητικά της ηλεκτρονικής πρόοδου. Καλώς, αν όλοι συμφωνείτε θα ψηφίσουμε διανατάσσεω της χειρός. Οπότε θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες ε, να το ελέγξουν και να κινητοποιηθεί και η γραμματεία για την καταμέτρηση. Ποιος είναι υπέρ της έκθεσης κυρίας Μπάουερ. Contre. Κατά. Qui s'abstient Apochette. 53... 53 ψήφισαν, 24 υπέρ, 29 κατά και καμία αποχή. Παρακαλώ, μείνετε στην αίθουσα. Θα επαναληφθεί η ψηφοφορία. Nous allons devoir recommencer le vote, car... Γιατί ψήφισαν 53. Δεν ξέρω αν συμμετείχαν και οι δύο επιπλέον του ΕΛΚ. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε 53 ψηφίσαντες, ενώ τα μέλη της Επιτροπής μας είναι 50. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Ε, Παρακαλώ. Οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων να ελέγξουν ότι τηρείται η ποσόστοση κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριο Ορή. Ναι. Εμεί είμαστε 18. Του μέτρησα. Συγγνώμη. Αλλά αυτό έπρεπε να το είχαμε κατάλαβει πριν, γιατί έφυγαν μερικοί, έφυγε ο κύριος Έλμερ, ε, ήταν πολύ γρήγορος. Με αφήστε τα παιχνίδια. Δεν παίζω κανένα παιχνίδι. Όταν η γραμματεία είπε ότι είμαστε 53, ε, αργήστε μέχρι να πείτε ότι κανονικά δικαιούμαστε να ψηφίσουμε μόνο 50. Και έφυγαν μερικοί. Δυστυχώς ε, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν λειτουργεί. Κύριε Ωρία, έχετε 18. Ας το ελέγξουν όλοι όλες οι ομάδες, παρακαλώ, σε ελέγξουν τα μέλη τους. Κύριε Κάζα, κύριε Σέρκας, έχετε 13 καταρχήν δικού σας. Κύριε Χάρκιν, έχετε 6 μέλη. Ε, πράσινοι. Τέσσερις δικαιούνται να ψηφίζουν πράσινοι ε, μεταρρυθμιστές ε, τρεις, γκουε τρεις, Ελευθερία και Δημοκρατία δύο, Ε, μη εγγεγραμμένους δεν είδα. Alors nous allons recommencer le vote. Ωραία. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ.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 Le vote euh, conduit à... Ψήφισαν 49, 24 υπέρ και 25 κατά, χωρίς αποχές. Συνάδελφοι, δεν έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη. Η έκβαση τη ψηφοφορία μα υποχρεώνει να καταθέσουμε νέα έκθεση επί της προτάσεως τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν λύσουμε όμω τη συνεδρίαση, έχουμε και άλλη μια ψηφοφορία για την εξέταση της γνωμοδότησης με τη μορφή επιστολής που θα στείλουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για την υπόθεση Nokia της Γερμανίας με αίτημα κινητοποίησης ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχετε λάβει την επιστολή. Ποιο είναι υπέρ του να στείλουμε επιστολή, γνωμοδότηση με τη μορφή επιστολή στην Επιτροπή Προπολογισμών. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα, οπότε ολοκληρώσαμε τις